Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, να αρχίσουμε σιγά σιγά την απογευματινή συνεδρίασή μας. May I welcome among ourselves, ε, Να καλωσορίσουμε τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Φρανς Τίμερμανς. Κύριε Τίμερμανς, είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιτέλους είστε εδώ στην Επιτροπή μας στο πλαίσιο αυτού του διαθεσμικού διαλόγου και θα θέλαμε να ανταλλάξουμε απόψεις για ζητήματα που μας απασχολούν όλους. Αναλογικότητα, επικουρικότητα, καλύτερη νομοθεσία. Προφανώς το έργο της Κομισιόν για τη δικαιοσύνη για τους καταναλωτές, την ισότητα των φύλων, τη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, τη συνεργασία, τις δικές σας απόψεις για την διοργανική συμφωνία διότι όπως γνωρίζετε η Επιτροπή μας είναι αρμόδια για την καλύτερη νομοθεσία, την εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας, της επικουρικότητας κτλ. Σημειώνω ότι έχετε περιορισμένο χρόνο και ότι θα πρέπει να φύγετε ακριβώς στις 4 Άρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση θα ήθελα να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκλησή σας. Ζητώ συγγνώμη για το γεγονός ότι χρειάστηκε να αναβάλουμε τη συνάντησή μας τον Οκτώβριο διότι ε, χρειάστηκε να πάω στην Τουρκία για να διαπραγματευτώ με τις τουρκικές αρχές το κοινό σχέδιο δράσης και σας ευχαριστώ για την κατανόηση που επιδείξατε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα και θα κάνω κάποια σύντομα σχόλια για να αφήσουμε περισσότερο χρόνο για τη συζήτησή μας. Τα σχόλιά μου αυτά θα επικεντρωθούν σε ορισμένα ζητήματα, κυρίως στην ε, διοργανική συμφωνία, στην οποία καταλήξαμε το Δεκέμβριο. Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Κομισιόν για την καλύτερη νομοθεσία. Και χαίρομαι πολύ που χαιρετίστηκε ε, την ε, προηγούμενη εβδομάδα στο, στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο κατά τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας και πρέπει να σας πω ότι τόσο οι αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με επικεφαλής τον Κίφερ Χόφσταντ όσο και η αντιπροσωπεία της Προεδρίας με επικεφαλής τον Νίκο Σμιτ επέδειξαν επικοδομητική στάση και εξευρέθη συμβαστική λύση στη βάση της πρότασης Κομισιόν και θα ήθελα να επισημάνω κάποια στοιχεία που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Πρώτα απ' όλα θα αυξήσουμε τη διαφάνεια του έργου μας δημοσιεύοντας τις προτάσεις μας σε πολύ πρώιμο στάδιο συμπεριλαμβάνοντας και μεγαλύτερο μέρος του παράγωγου δικαίου έχουμε αποσαφηνίσει το ζήτημα των εκτελεστικών και κατεξοδότηση πράξεων που ήταν ένα ζήτημα που συζητήθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου περισσότερο από ό,τι με την Κομισιόν σε κάθε περίπτωση σημειώθηκε κάποια πρόοδος αλλά πλέον ε, το ζήτημα αυτό αφορά κυρίως αυτά τα δύο όργανα δημιουργήσαμε την ε, δυνατότητα με τον τρόπο που οργανώσαμε την ε, διαδικασία refit εκ παραλίλου με το ετήσιο, ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν να υπάρχει και μια κατάρτιση του προγράμματος REFIT, κάτι που θα μας επιτρέψει να, να συζητούμε για το ποιοι τομείς θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο και τι θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση για τη μείωση της γραφειοκρατίας, για τον εξυγχρονισμό ή για τον εξορθολογισμό ορισμένων νομοθετημάτων και με αυτόν τον τρόπο να απαλλαγούμε από παροχημένη νομοθεσία που εξακολουθεί να ισχύει. Θεωρώ ότι αυτό για το Κοινοβούλιο μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο όχι μόνο για τη θέσπιση νέας νομοθεσίας αλλά και για... Ε, μια εκαθάριση, να το πω έτσι, της ισχύουσας νομοθεσίας και υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Να τονίσω επίσης στο πλαίσιο αυτό ότι κανένα από τα θεσμικά όργανα δεν αμφισβήτησε το γεγονός ότι μιλούμε για καλύτερη νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση δεν μιλούμε για χαμηλότερες φιλοδοξίες ή ε, επιδείνωση της ποιότητας. Αντιθέτως, διατηρούμε τα πρότυπα ποιότητας, αλλά με λιγότερο βάρος, με λιγότερο, μικρότερο φόρτο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επίσης θα ήθελα να χαιρετήσω την ενεργό ε, δραστηριότητα της ε, Επιτροπής σας για μια σειρά αποζητήματα, λογοδοσία, διαφάνεια, ε, λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και σας διαβεβαιώ ότι όλα αυτά τα θέματα θα αποτελέσουν αντικείμενο του θεματολογίου για την καλύτερη νομοθεσία. Αυτά για να αφήσω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε για τις εισαγωγικές σας αυτές παρατηρήσεις. Ο κύριος Χρυσόγονος έχει ζητήσει το λόγο πρώτος. And uh, welcome, Mr. Vice President. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Πριν από δύο μέρες το ελεγκτικό συνέδριο δημοσίευσε τα απορίσματά του για τα πέντε προγράμματα διάσωσης για υπερχρεωμένα κράτη-μέλη. Και τα πορίσματα αυτά αποκαλύπτουν ότι υπήρξαν ανισότητες στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη ε, δέχτηκαν ε, την συνδρομή της Κομισιόν στη διάρκεια αυτών των προγραμμάτων διάσωσης και ότι θα πρέπει να αντιληφθούν σοβαρά διδάγματα όσον αφορά τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων από την πλευρά της Κομισιόν. Επομένως θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ε, αποδέχεστε τα απορίσματα αυτά του ελεγκτικού συνεδρίου και αν υπάρχει, αν έχετε προγραμματίσει κάποια διαδικασία προκειμένου να διαπιστώσετε ποια ήταν τα λάθη που έγιναν και πώς θα μπορούσε να υπάρξει στο μέλλον καλύτερη διαχείριση όταν θα αντιμετωπίζουμε παρόμοιες καταστάσεις. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αλλά δεν μπορώ να απαντήσω ακόμα. Αυτή η έκθεση ε, δημοσιεύτηκε προχτές Βεβαίω θα λάβουμε υπόψη μας πλήρως ε, την έκθεση, αλλά δεν είχαμε ακόμα καν τη δυνατότητα να ενημερωθούμε, να τη διαβάσουμε. Επομένω δεν μπορώ επισήμως να ανταποκριθώ ε, στα ευρήματα, στις παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να σα διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα ε, αντιδράσει, θα απαντήσει, όπως πάντα το κάνει στις εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου και υποθέτω κιόλα ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντήσει θα μπορούσαμε στην ε, κοινοβουλευτική σα επιτροπή ή και σε άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ να συζητήσουμε και τα πορίσματα του Ελεκτικού συνεδρίου και την απάντηση τη επιτροπή. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σα πω τίποτα περισσότερο. Ο λόγο ύπαρξη του ελεγκτικού συνεδρίου είναι να αντλούμε διδάγματα από τα πορίσματά του. Επομένω, ευχαρίστω να τα συζητήσουμε αυτά τα διδάγματα κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε, κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, κύριε Τίμερμαν. Δύο ερωτήσεις. Το ένα αφορά την συμμετοχή των πολιτών. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι μας είπατε ότι θα αυξήσετε τη διαφάνεια ε, της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων ώστε να διασφαλίσετε και έναν δημόσιο έλεγχο στο διαδίκτυο από πλευράς πολιτών. Για μας αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Εγώ είμαι η συγγήτρια της ετήσιας έκθεσης για τη δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων από πολίτες και από τα σχόλια ε, τα οποία διάβασα κατά τη ε, ε, διαβούλευσή μου με τους πολίτες και με την κοινωνία των πολιτών, φαίνεται ότι πολύ συχνά υπάρχει έλλειψη συμμετοχής. Ενώ είναι διαθέσιμα τα έγγραφα, πολύ δύσκολα μπορεί να τα κατανοήσει κανείς. Επομένως, θα έπρεπε ίσως να προσπαθήσουμε να αξιολογούμε το ενδεχόμενο να υπάρχει μια μορφή ε, πιο ευανάγνωστων κειμένων υπό την έννοια ότι θα πρέπει να γίνονται καλύτερα αντιληπτά, να υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος επικοινωνίας, ώστε να να αντιληφθούν ακριβώς οι πολίτες τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά φυσικά και στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Υπάρχουν ε, κάποια ζητήματα τα οποία είναι πολύ πιο εύκολα στην επικοινωνία τους, ε, κάποια άλλα που είναι πιο δυσνόητα βέβαια για τους πολίτες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε τη συμμετοχική δημοκρατία, κάτι ή μάλλον αυτό που αρέσει πιο πολύ σε εμά την αμεσοδημοκρατία. Ε, σε σχέση με τους πολίτες. Και ε, κάτι άλλο σημαντικό αφορά του τριμερείς διαλόγους. Το συζητούμε πολύ το θέμα των τριμερών διαλόγων, διότι αφενός θεωρούμε ότι πρέπει να εγγυηθούμε και να προστατεύσουμε ε, αυτή τη διαδικασία λήψης απόφασης και το πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το στάδιο, διότι είναι το στάδιο της διαπραγμάτευσης, αλλά αφετέρου πρέπει να διασφαλίσουμε και διαφάνεια με ε, αυτής της τόσο σημαντικής ε, φάσης της διαδικασίας που ακόμα ε, δεν υπάρχει και προσπαθούμε να δούμε με τους συναδέλφους πώς θα πρέπει να του ορίσουμε αυτούς τους τριμερείς διαλόγους. Είναι ένας χώρος περισυλλογής, space to think ή ένας χώρος για να αποφασίσουμε, space to decide. Εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις λοιπόν. Σας ρωτώ τι άποψη έχετε λοιπόν προκειμένου να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και για τους τριμερείς διαλόγους, τις διαπραγματεύσεις δηλαδή μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Σας ευχαριστώ πολύ. Δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι το να αναρτήσει κάποιο ένα έγγραφο, μια πρόταση, μια ιδέα δημοσίω κάπου, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει μεγαλύτερη ε, συμμετοχή του κοινού. Πολλά από αυτά τα οποία καταρτίζουμε είναι τεχνικά περίπλοκα, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε καν εμείς, ε, όχι τώρα το ευρύ Δεδομένων και των εγγράφων τα οποία ε, δημοσιεύουν τα θεσμικά όργανα, είναι αδύνατο να γίνει μια δημόσια μετάφραση, αν θέλετε, όλων των εγγράφων που δημοσιεύονται. Ε, θα επιβαρύνει πάρα πολύ ε, εμάς και δεν έχουμε και τέτοιες δυνατότητες. Αυτό που μου αρέσει να σκέφτομαι είναι ότι αυτή τη στιγμή ε, ξεκινήσουν τα πάντα και δημοσιευτούν εντός 8 ή 12 εβδομάδων δημοσίως υπάρχουν ε, αρκετοί ε, και συγκεκριμένοι ιδιώτες αλλά και οργανώσεις που ενδιαφέρονται άμεσα για κάποιο ζήτημα. Εγώ θα ήθελα, ίσως σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από κάποιο διάστημα, αυτές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή αυτοί οι ιδιώτες να ε, μας πούν ποια είναι η εμπειρία τους με αυτό το νέο τρόπο εργασίας και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε ίσως θα μπορούσαμε ίσως να το θέσουμε και ως θέμα συζήτηση στην πλατφόρμα του το που εχουμε έχουμε κράτη-μέλη και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών επίσης. Θέλω λοιπόν να βελτιωθεί η διαδικασία, αλλά θα ήθελα να αντιληφθείτε ότι ε, άμεσα είναι λίγο περιορισμένα αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει όμως και ε, βοήθεια που μπορούμε να λάβουμε από τους πολίτες να μας πούν την άποψή τους απευθείας ε, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και με τη δική σας την Επιτροπή και με άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου ώστε να την υλοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Διότι συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί σας ότι αν θέλουμε πραγματικά να ασχοληθούν περισσότεροι οι πολίτες με αυτά που κάνουμε πρέπει να κατανοήσουν και τι κάνουμε. Ε, και πολλά από αυτά που κάνουμε είναι ιδιαίτερως τεχνικά. Κάποιο αγοράζει ένα αυτοκίνητο όχι για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κινητήρα, αλλά για τη συμπεριφορά του στο δόστρωμα. Ε, ο κόσμο ε, αποδέχεται την νομοθεσία όταν είναι αποτελεσματική, κάνει αυτό για το οποίο έχει εκπονηθεί και όταν δεν είναι αποτελεσματική, όταν δεν κάνει αρκετά, την απορρίπτει. Πρέπει λοιπόν να γίνει ένα διάλογο από αυτού και ελπίζω να έχουμε και απαντήσει από του πολίτε όταν θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Όσον αφορά του τριμερεί διαλόγου. Η οδυνηρή μου εμπειρία με έχει διδάξει ότι πρέπει να προσέχω πάρα πολύ τι λέω για τους τριμερείς διαλόγους. Διότι στο παρελθόν ε, ασχολούμαν με, το κοινοβουλευτικό, ε, με τον κοινοβουλευτισμό και ε, κάθε φορά που προσπαθούσα να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα ε, βρισκόμουν ζημιωμένος και πάντα μου λέγανε ότι δεν είναι δική σου δουλειά αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω λοιπόν να μπω σε αυτά τα σκοτεινά μονοπάτια, μεν, αλλά από την άλλη δεν μπορώ και να συγκρατηθώ. θα μπορούσατε ίσως κατά περίπτωση να, πρόταση αυτή να χρησιμοποιήσετε τον πλήρη νομοθετικό κύκλο που είναι διαθέσιμος για τους συνομοθέτες βάσει των συνθηκών. Δεν είναι απαραίτητο να ε, καταφεύγουμε πάντα στον τριμερή διάλογο ως λύση. Ε, αυτή είναι η ταπεινή άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Πράγματι ενδιαφέρουσα η πρότασή σας για τον τριμερή διάλογο, αλλά εγώ θα ήθελα να μιλήσω για κάτι το οποίο ίσως ε, μπορείτε να συζητήσετε πιο άνετα, τη διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. τα πρώτα βήματά σας ήταν ενθαρρυντικά πέρσι, Το Δεκέμβριο του 2014 ξεκίνησε η δημοσίευση των συνεδριάσεων των ομάδων πίεσης των πιο σημαντικών ομάδων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έκτοτα ε, όμως υπήρξαν αρκετά ερωτηματικά για το κατά πόσο είναι χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες, εάν ε, ε, ίσως τα πιο τεχνικά γίνονται σε επίπεδο εργασίας και σε διοικητικό επίπεδο στις γενικές διευθύνσεις. Και ερώτησή μου λοιπόν είναι αν όντω πρόκειται για το πρώτο βήμα προς μεγαλύτερη διαφάνεια, μέχρι πού έχουμε φτάσει, ε, αν μπορούμε πραγματικά να έχουμε μια πλήρη στρατηγική από όλα τα θεσμικά όργανα όσον αφορά την ε, συμπεριφορά προς τους ομάδες πίεσης, προς τα λόμπι και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και στις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Θα ήθελα να αναφέρω και ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έχει ε, προκαλέσει πονακεφάλους και στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το θέμα των γραπτών ερωτήσεων ε, των Ευρωβουλευτών. Αφενός φαίνεται να υπάρχει μια ενόχληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον αριθμό των ερωτήσεων και για το χρόνο που χρειάζονται για να απαντήσουν ε, σε αυτές τις ερωτήσεις και από την άλλη, από την εμπειρία μου ως Ευρωβουλευτής, εγώ έχω θέσει περίπου 20 ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της θητείας και δύο εξ αυτών των ερωτήσεων απαντήθηκαν σχεδόν εγκαίρως, όλες οι υπόλοιπες ε, ήταν πέραν των ε, διοριών που προτείνονται και φυσικά η ποιότητα των απαντήσεων πολύ συχνά ήταν ε, ε κάτι σαν δελτίο τύπου ε, ε, που θα δίναμε σε ένα δημοσιογράφο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλές φορές πήρα πολύ περισσότερες πληροφορίες από το ε, για το θέμα για το οποίο ρωτούσα, θέτοντα απλώς ερώτηση ε, ως απλός πολίτης ε, μέσω της ε, ε, δυνατότητας αυτής της ελευθερίας ενημέρωσης. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε ε, στα πλαίσια του διαλόγου και της λογοδοσίας. Φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο δεν λαμβάνεται και τόσο σοβαρά και το χρησιμοποιείτε μόνο για στατιστικούς λόγους. Διαφάνεια. Καταρχάς ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για να ε, κατοχυρώσουμε θεσμικά τη διαφάνεια. Ε, θα εξυπηρετούσε και εμένα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε αυτό που κάνει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι οι ευρωβουλευτές δημοσίευσαν όλες τις συνεδριάσεις που κάνουν, να υπάρχει ένα μητρό σαν το δικό μας. Ε, αυτό θα ενισχύσει και όλους εμάς που θέλουμε να προχωρήσουμε το θέμα έτσι περαιτέρω. Αυτό το οποίο δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα είναι όταν το Κοινοβούλιο ε, προσπαθεί να ρίξει το βάρος μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε ότι η Επιτροπή πρέπει να κάνει αυτό και εκείνο και το άλλο και εμείς επειδή είμαστε αιρετοί δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Εγώ δεν το δέχομαι. Έχω εκλεγεί έξι φορές στο Εθνικό Κοινοβούλιο και ακόμα ε, θεωρώ ότι τα έγγραφά μου είναι δημόσια και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αμφιλεγόμενο επ' αυτού. Ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λοιπόν από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ίσως να πείσουμε και το Συμβούλιο να προχωρήσει λίγο επί του ζητήματο, ε, που είναι ίσως και η πιο τρομακτική εκ των προκλήσεων. Τώρα, το ερώτημα του σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να εργαζόμαστε. Έχω πει επανειλημμένω ότι εγώ είμαι ανοιχτό και θέλω να δω τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Πρέπει όμω να παραδεχτώ ότι υπάρχουν και κάποια όρια και ότι κάποιοι αξιωματούχοι έχουν συνεδριάσεις ε, μεν, αλλά δεν ε, ε, λαμβάνουν αποφάσεις και δεν έχουν και εξουσιοδότηση να λάβουν αποφάσεις. Αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις πρέπει να ε, λογοδοτούν απόλυτα για το τι λένε. Παραδείγματο χάρη, αν είσαι διευθυντής, επικεφαλής μιας οργάνωσης, πρέπει να προστατεύεις και τους ανθρώπους της οργάνωση, του οργανισμού σου, που δεν μπορούν να ε, προστατεύσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Αλλά όπως σας είπα, είμαι διατεθειμένος να να τα δούμε και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ταυτόχρονα όμως ε, νιώθω και μια ευθύνη ότι πρέπει να προστατεύσω τους ανθρώπους που εργάζονται για μένα και που δεν βρίσκονται στο ιεραρχικό επίπεδο ε, στο οποίο θα πρέπει να λογοδοτούν όταν δεν είναι αυτοί υπεύθυνοι για να λάβουν αποφάσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει δέουσα ισορροπία εκεί. Στο κάτω-κάτω της γραφής, εάν ακολουθείς μια γραμμική λογική, ο πιο νεαρός ε, ασκούμενος ε, θα ήταν υποχρεωμένος ε, να δημοσιεύει το πρόγραμμά του. εκεί μετά ξεκινάμε μια διαδικασία χωρίς τέλος. Πρέπει να είμαστε λίγο λογικοί, να γίνει μια συζήτηση επ' αυτού. Δεν λέω σε καμία περίπτωση, αλλά πρέπει να γίνει μια συζήτηση στα πλαίσια της ευρύτερης συζήτησης που πρέπει να γίνει και να υπάρξει, ελπίζω, μια διοργανική συμφωνία. Όσον αφορά τις γραπτές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ που φύγετε και πάλι το ζήτημα. Νομίζω ότι φέτος ε, είμαστε λίγο καλύτερα. Προλαβαίνουμε και τις διορίες. Ε, πίεσα λίγο για να είμαστε λίγο καλύτεροι σε αυτό. Να απαντάμε γέρος. Αλλά εδώ θα σας προκαλέσω λίγο εγώ από την πείρα που έχω αποκομίσει και ως εθνικός βουλευτής. Κάποιες φορές ως εθνικός βουλευτής μας ενδιαφέρει περισσότερο να θέσουμε την ερώτηση και όχι να περιμένουμε την απάντηση. Αυτό που βοηθά ώστε να επικεντρωθεί ε, μια διοίκηση ε, είναι να κάνετε περωτήσει αν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική. Ε, αυτό έκανα εγώ ως εθνικός βουλευτής. Αν πίστευα ότι μου έδιναν μια αμφίσιμη απάντηση ή δεν μου απαντούσαν πραγματικά, τότε έκανα μια δεύτερη ερώτηση. Και αυτό το έχω δει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους συναδέλφους. Ε, μεγαλύτερο επίπεδο ε, λεπτομέρειας και προσοχής, διότι φαίνεται ότι το Κοινοβούλιο αρχίζει να δαγκώνει λίγο περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Επομένως πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και πρέπει να είμαστε όλοι σε παγρύπνηση. Αυτό νομίζω ότι είναι η σύστασή μας, να τους έχετε σε παγρύπνηση είναι και μια διαδικασία την οποία όλοι διδασκόμαστε κάποια πράγματα. Εμείς θέλουμε να είμαστε πιο ανοιχτοί και να σας απαντούμε πλήρως αυτό που θέλετε. Μπορεί να μην είναι απάντηση που, που περιμένετε, αλλά θα πρέπει να είναι πλήρης απάντηση στην ερώτησή σας. Εγώ έχω βρεθεί και από τις δύο πλευρές της κυβέρνησης, έχω βρεθεί και στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση και ξέρω ότι αυτό δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε εθνικότητα ή δεν είναι θέμα νοοτροπίας λαού. Ε, όλοι θέτουμε ερωτήσεις και χρειαζόμαστε απαντήσεις ε, και... Ε, πραγματικά είμαι διατεθειμένος να συνεργαστούμε και να υπάρξει και διάλογος με, εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι έγιναν κάποια θετικά βήματα την περασμένη χρονιά ή τουλάχιστον έτσι ελπίζω. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ το γεγονός που παρά το πολύ φορτωμένο πρόγραμμά σας βρήκατε χρόνο για να έρθετε εδώ. Θέλαμε λοιπόν να, ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας, να σας πούμε τα δικά μας σχόλια. βήμα προς βήμα προσεγγίζουμε στον στόχο της καλύτερης νομοθεσίας. Νομίζω ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να διδαχθούν το ένα από το άλλο και να προσπαθήσουν να προσαρμόσουν τους μηχανισμούς, τα μέσα και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν για να βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Να αναφερθώ εγώ στην, ε, στις προφορικές ερωτήσεις. Όντως η Γιουλιάνε Ρέντερ έχει και Ορισμένες φορές οι ε, απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές. Τα παλαιότερα χρόνια όταν τίθεντο ε, ερωτήσεις φάνηκε κάποια στιγμή ότι πρόκειται για μια διαδικασία από συγκεκριμένα μέλη τα οποία δεν ήταν ιδιαίτερα δραστήρια ε, κατά τα άλλα ε, έρχονταν και έθεταν προφορικές ερωτήσεις σαν να το κάναν ε, κατά κάποιο τρόπο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και για μεγαλύτερη προσοχή. Και πολλές φορές δεν ήταν ιδιαίτερα καλές οι ερωτήσεις. Άρα αν οι ερωτήσεις που θέτουμε είναι καλές, καλές θα είναι και οι απαντήσεις. Για τη διαφάνεια φυσικά είναι ζητούμενο. Ωστόσο, όταν συζητούμε το ενδιαφέρον που ενδεχομένως να επιδείξει η κοινή γνώμη για την ε, αναθεώρηση της ε, νομοθετικής διαδικασίας, ε, μάλλον δεν θα επιδειχθεί και ιδιαίτερο ε, ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Ωστόσο, η διαφάνεια είναι κρίσιμα σημασία γιατί δεν αφορά μόνο τη δημοσίευση συγκεκριμένων πληροφοριών αλλά και την αποφυγή συγκεκριμένων λαθών εκ μέρου τη Κομισιόν. Α είμαστε ειλικρινεί. Υπήρξαν κάποιες ανόητε θα έλεγα ε, νομοθετικέ πρωτοβουλίες στο παρελθόν οι οποίες ε, ε, δημιούργησαν και κάποια γελιοποίηση στα ευρωπαϊκά όργανα. Και ας είμαστε ειλικρινεί. αυτά τα σφάλματα δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Ε, μιλώ για κάτι λιθιότες όπως εκείνες με τις, ε, με, το, με τις μπανάνες και το σχήμα των αγκουριών και και κάποιε άλλες πρωτοβουλίες που εν πάση περιπτώσει δεν ε, στέφθηκαν και με ιδιαίτερη επιτυχία. Σε κάθε περίπτωση στόχος όλων μας είναι η καλύτερη νομοθεσία που θα αποβαίνει σε όφελος όλων και των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δημοσιεύονται, να δημοσιεύονται τα πάντα, ιδιαίτερα όσον αφορά τους ε, τριμερείς διαλόγους. Και σε αυτό το θέμα συμφωνώ με τον Πρόεδρο η ανταλλαγή απόψεων στη διαδικασία ε, ε, που ακολουθείτε δεν θα πρέπει να ξεκινά στο στάδιο του τριμερούς διαλόγου. Θα πρέπει πριν από τον τρίμερο, τριμερή διάλογο να δημοσιεύονται συγκεκριμένες πληροφορίες. Κάτι που θα καταστήσει και τον ίδιο τον τριμερή διάλογο πιο αποτελεσματικό. Γνωρίζουμε μια και μιλώ για τον ε, τριμερή διάλογο, ότι υπάρχουν διάφορα τρίκ και διάφορες ε, διαπραγματευτικέ στρατηγικές που ακολουθούνται. Ενδεχομένως, η δημοσίευση τέτοιων ε, πληροφοριών να μην αποβεί σε όφελος των θεσμικών ε, οργάνων. Για μένα το κυριότερο είναι η αποτελεσματικότητα των νομικών πράξεων και σε δεύτερη μοίρα μπαίνει η διαφάνεια. Οι νομικές πράξεις θα πρέπει να γίνονται σεβαστές, να γίνονται κατανοητές και να εφαρμόζονται. Και τέλος δύο ερωτήματα θα ήθελα να σας ε, θέσω. Χαιρετίζω το γεγονός ότι η καλύτερη νομοθεσία είναι στόχος αναγκαίος για να δοθεί μια τόνωση στην οικονομία, να ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης κτλ. κτλ. Είναι η μοναδική μας δυνατότητα να ενισχύσουμε την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη σημασία η καλύτερη νομοθεσία. Ωστόσο, νιώθω ότι υπάρχει μια έλλειψη, μια απουσία που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσον αφορά τη διαθεσμική ε, συμφωνία. Αλλά ελπίζω ότι θα συμπεριλάβετε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στη συμφωνία αυτή στο άμεσο μέλλον. Και τέλος, αξιολόγηση επιπτώσεων. Οι αξιολογήσει επιπτώσεων θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο που θα μα επιτρέπουν να αποφεύγουμε σφάλματα με σκοπό την θέσπιση καλύτερη νομοθεσία. Ιδίω όταν πολλέ φορέ η διαδικασία νομοθέτηση διαρκεί ε, τρία ε, χρόνια ή και περισσότερα. Πολλές φορές η πραγματικότητα αλλάζει όταν ξεκινά να, να ένα νόμο το 2016 και τελειώνει το 2020, ενδεχομένω τα πρακτικά στοιχεία, η πραγματικότητα ίδια να έχει αλλάξει. Τώρα το ερώτημά μου. Όσον αφορά τα μέσα και τους μηχανισμούς που προβλέπονται σε αυτή τη συμφωνία, ελπίζω να έχουν ληφθεί υπόψη δύο διαστάσεις. Η, η ανάπτυξη της οικονομίας και η ρεαλιστική αξιολόγηση των επιπτώσεων των νομικών πράξεων. Ελπίζω αυτά τα δύο στοιχεία να έχουν τονιστεί στην συμφωνία με τον τρόπο που έχουμε περιγράψει εμείς. Ευχαριστώ. Εσείς ε, αναφερθήκατε στις συγκεκριμένε ερωτήσεις. Εγώ ποτέ δεν θα σχολίαζα την ποιότητα, το επίπεδο ερωτήσεων ευρωβουλευτών. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ε, μπορούμε όντως σε ορισμένες περιπτώσεις να βελτιώσουμε τις δικές μας απαντήσεις σε κάποιες ε, απαντήσεις όντως ενδεχομένως να είναι λίγο, λίγο και με μια διακριτικότητα προκλητική η απάντηση της Κομισιόν. Ε, έχει γίνει αυτό στο παρελθόν, γι' αυτό και εγώ δεσμεύομαι ότι σε στενή συνεργασία μαζί σας θα βελτιωθούμε, ιδιαίτερα όσον αφορά την έγκαιρη απάντηση στα ερωτήματά σας. Επίσης συμφωνώ ότι στην νομοθεσία κάνουμε κάποιες φορές ηλίθια λάθη. Μπορεί κανείς να χάσει μέχρι και εκλογές για κάποιο ίσονο σημασία ζήτημα. Και ενδεχομένως κάποιες φορές κάτι που πραγματικά έχει νόημα και είναι σημαντικό για μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, στο ευρύ κοινό να φαίνεται γελίο. Άρα, το να βάλεις ένα τέτοιο στοιχείο στο ίντερνετ σε πολύ πρώιμο στάδιο, διαδρέχει τον κίνδυνο να το διαβάσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κοινή λογική και οι οποίοι μπορεί να αναρωτηθούν καλά είναι δυνατόν τώρα αυτοί νομοθετούν για, για το σχήμα των μπουκαλιών λαδιού που θα έχουν στα τραπέζια τους στα εστιατόρια. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Κάποιες φορές δε ε, έχω την αίσθηση ότι κάποιοι ευρωβουλευτές μας ασκούν άδικη κριτική. το ζήτημα, αναφέρομαι στο ζήτημα με τα κεριά. Υπήρξε ε, μια περίπτωση όπου αναφέρθηκε στην Κομισιόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αποκλίνοντες ε, κανόνες ε, και πρέπει να δημιουργηθούν ενιαίοι κανόνες για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά μας. Και μας ζητήθηκε να συντάξουμε έναν συγκεκριμένο κανόνα για τα κεριά ώστε να ισχύσει σε όλη την ενιαία αγορά. Εμείς ε, στη συνέχεια το ψάξαμε το θέμα και ανταποκριθήκαμε σε αυτό το αίτημα της βιομηχανίας και των κρατών μελών και στη συνέχεια από τα 28 κράτη-μέλη τα 27 υποστήριζαν αυτήν την πρόταση που υποβάλαμε και μία χώρα απήχε από την ψηφοφορία. Και ξαφνικά εμφανίζεται στις εφημερίδες ότι αυτοί οι ηλίθιοι τύποι στην Κομισιόν θέλουν να ρυθμίσουν μέχρι και το ζήτημα του σχήματος των ε, ε, κεριών. Εδώ είχαμε όμως μια, ένα παράδειγμα καλύτερης νομοθεσίας. Αντί να ε, έχουμε 28 κράτη-μέλη και αντίστοιχες εθνικές οικονομίες και εθνικές βιομηχανίες να προσπαθούν η καθεμιά για τον εαυτό της να επιβιώσει, θεσπίσαμε κανόνες κοινούς, ενιαίους, οι οποίοι θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και σε δεύτερο χρόνο θα αυξήσουν και τις θέσεις απασχόλησης. Ωραία, οπότε εγώ λέω, κάποιες φορές κάνουμε ανόητα σφάλματα, αλλά κάποιες φορές, κάποιες άλλες φορές, ε, ζητήματα που σχετίζονται με την καλύτερη νομοθεσία δέχεται να παρουσιάζονται ως ε, ανόητα σφάλματα. Ε, αναφερθήκατε στον τριμερή διάλογο και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχει πάντοτε η ανάγκη να εξευρίσκεται μια ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια. Εγώ είμαι πάντοτε υπέρ της διαφάνειας ακόμα και σε ζητήματα που ε, είναι αμφισβητήσιμο το αν η διαφάνεια προσθέτει το Αλλά πάντοτε εγώ θεωρώ ότι έχει σημασία να υπάρχει διαφάνεια. Πολλές φορές η νομοθεσία είναι δυσνόητη ή και ακατανόητη ε, στους ε, απλούς πολίτες, αλλά παρόλα αυτά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να δημοσιεύονται τα έγγραφα. Όποτε έχει κανείς αμφιβολία, εγώ θεωρώ ότι η λύση είναι η ενίσχυση της διαφάνειας. Βεβαίως όχι με τρόπο που να εμποδίζει το έργο μας. Και συμφωνώ μαζί σας ότι ορισμένες φορές η αμοιβαία εμπιστοσύνη μπορεί να βοηθά τους ανθρώπους ε, να ε, ε, βρίσκουν λύσεις χωρίς να εκτίθενται σε όλη τη διαδικασία μιας διαπραγμάτευσης στη δημόσια σφαίρα. Ε, αυτό ε, είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι οι πολιτικοί. Για τον έλεγχο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι αν κάνουμε τη δουλειά μας σωστά στην πλατφόρμα Refit, χωρίς να το αποκαλέσουμε τεστ ε, έλεγχο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα επιτύχουμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα αυτά που ζητάτε κι εσείς. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι καν ε, πολιτικά χρωματισμένο ζήτημα. Καταλαβαίνω ποια είναι η θέση σας. Έχουμε συζητήσει άλλο το θέμα, άλλωστε το θέμα και άλλες φορές. Για την ε, μελέτη επιπτώσεων. Εγώ θα ήθελα να πάμε και πιο πέρα, αλλά μέχρι εκεί καταφέραμε να φτάσουμε ε, σύμφωνα με τη Διοργανική Συμφωνία και σίγουρα αποτελεί μία ε, πρόοδο το Συμβούλιο Διοικητικού Ελέγχου, Ρυθμιστικού Ελέγχου ε, θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από εδώ και στο εξή. Θα υπάρχουν και τρία ανεξάρτητα εξωτερικά ε, μέλη. Εγώ μάλιστα θα πρότεινα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και ε, άτομα που ενδεχομένως να εργάζονται για άλλα θεσμικά όργανα. Προς το παρόν όμως, εγώ θα, το έβρισκα ως μια θετική εξέλιξη στο μέλλον. Προς το παρόν όμως, σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως ε, θεσπίστηκε το όργανο αυτό, θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, ε, θα είναι πολύ πιο επικριτική η στάση του οργάνου απέναντι στις δικές μας προτάσεις Θεωρώ ότι θα κάνει πολύ διεξοδικότερη δουλειά από ότι στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας τρόπος ε, να ελέγχεται με ταχύ τρόπο ε, μια διαδικασία refit, ε, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες. Γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές μπορεί να προσπαθήσεις να ε, σχεδιάσεις άλογο και να σου βγει καμήλα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ε, εξετάζεται η επίπτωση μιας μεγάλης ε, τροποποίησης αν υπάρχει. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα τέταρτο, 13 λεπτά και τέσσερις ομιλητές. Με την άδειά σας λοιπόν θα δεχτώ και τις τέσσερις ερωτήσεις μαζί ώστε να μπορέσετε τουλάχιστον να, να απαντήσετε έστω και λίγο. Καταρχάς, ο κύριος Κέστερ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της διαφάνειας όπως και η Λάρα Φεράρα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, συμφωνίες ε, εμπορικών συναλλαγών, ΣΥΤΑ και TTIP. Ποια ήταν η συμπεριφορά της Κομισιόν απέναντι στους ευρωβουλευτές. Πριν από 1,5 χρόνο όταν εξελέγην, ε, έθεσα ερώτημα στην Κομισιόν για ποιο λόγο δεν έχω πρόσβαση στα έγγραφα. Και μου απάντησαν λακωνικά ότι η διαπραγμάτευση αυτή γίνεται εμπιστευτικά και ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Θα θέσω τώρα το ερώτημα και ας ακουστεί κάπως ανόητο. Αυτό ήταν ένας τρόπος ενίσχυσης της αδιαφάνειας. Επίσης, αφήνεται να δημιουργούνται διάφορες ασάφειες και να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα. Γι' αυτό εγώ ως ευρωβουλευτής θεωρώ ότι θα έπρεπε οι διαπραγματεύσεις για το TTIP και το ΣΥΤΑ να χαρακτηρίζονται από περισσότερη και μεγαλύτερη διαφάνεια. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και το αναγνωρίζω αυτό, αλλά θα ήθελα ε, με βάση ε, την, ε, θα ήθελα να αναφερθώ ε, στη δυνατότητα να διαβάσει κανείς ορισμένα έγγραφα μπορεί να κρατήσει και κάποιες σημειώσει αν θέλει, χωρίς να του παραδίδονται, αλλά γνωρίζετε ότι είναι πολύ περίπλοκα τα θέματα αυτά ε, και πολλές φορές δεν αρκεί να διαβάσει τόσο περίπλοκο έγγραφο μόνο μία φορά. Και έτσι δεν έχουμε τελικά τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε μια συνολική εικόνα για τις διαπραγματεύσεις που γίνονται για αυτές τις συμφωνίες εμπορίου. Και όταν μάλιστα καλούμε να υπογράψω και κάποια δήλωση ασφαλείας σύμφωνα με την οποία δεσμεύομαι ότι ε, τα θέματα που, διάβασα και τις πληροφορίες που διάβασα δεν μπορώ να τις ανακοινώσω στους ε, ψηφοφόρους μου ή στους πολίτες της ε, εκλογικής μου ε, περιφέρειας γιατί αυτό θα ήταν ποινικά κολάσιμο αυτό δεν είναι κάτι που συνάδει με την αρχή της διαφάνειας. Οπότε το ερώτημά μου είναι τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου να ενισχύσετε τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις για τις εμπορικές συμφωνίες αυτές και τι θα κάνετε προκειμένου εμείς οι ευρωβουλευτές να μπορούμε και στις εκλογικές μας περιφέρειες να ε, συζητούμε για τα θέματα αυτά με τους ψηφοφόρους μας. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους, τους συναδέλφους που θα πάρουν μετά το λόγο να περιορίζονται στο χρόνο που τους αναλογεί για να μείνει χρόνος και για τις απαντήσεις. Κύριε Χάουταλα. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, σήμερα το πρωί φτάσαμε σε ένα σημαντικό βήμα, σε μια πορεία την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ακολουθήσει εδώ και πολλά χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια. Ε, έχω την τιμή να είμαι εισηγήτρια για το θέμα αυτό είναι ο προτινόμενος κανονισμός για την διοικητική διαδικασία. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και με την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα της Επιτροπής, την κυρία Μίχου, και ο κύριος Λεγκάλ από την νομική υπηρεσία του ε, Συμβουλίου ε, μας απάντησε και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Αυτό που με εντυπωσίασε αρνητικά ή μάλλον θετικά, είναι ότι κανείς δεν μας είπε κατευθείαν όχι. Νομίζω θα ήταν καλύτερα, θα ήταν πολύ καλύτερο για την δική σας ε, διαδικασία του ευνομοθετήν να μην απορρίψετε ε, εκ προημίου αυτή την ε, πρόταση για τη βελτίωση της διοικητικής διαδικασίας. Πολλοί εμπολιτές, ανάμεσά του και ο πρώην διαμεσολαβητής κ. Διαμαντούρο, είπαν ότι ένα τέτοιο κανονισμό για την δημόσια για τη διοίκηση, την ευρωπαϊκή διοίκηση, θα μπορούσε να διευκολύνει και τη δική σα ζωή, θα μπορούσε να διευκολύνει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν μαζί της πολίτε και ε, οργανώσει. Ε, μας επεσήμανε επίσης ο κύριος Διαμαντούρο ότι ε, όταν ξεκίνησε τη θητεία του ε, είχε ε, να ασχοληθεί με τέσσερι υπηρεσίε τη Επιτροπή, ενώ τώρα έχουμε φτάσει στι 64 και πολλές από αυτές ακολουθούν τους δικούς τους κανόνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πλήττει και την βιομηχανία και τις ε, επιχειρήσεις. Επομένως θεωρώ ότι με όλα αυτά κάποια στιγμή θα φτάσουμε να σας πείσουμε για την ανάγκη αυτού του κανονισμού. Κυρία Γοζιέ, ευχαριστώ. Χαίρομαι που άκουσα την παρουσίαση των στόχων που έχετε εσείς και πώς βλέπετε το ζήτημα ε, για την ε, στην ε, συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Υπάρχει το ζήτημα του πώς πού στέκεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε όσα είναι απαραίτητα, αλλά χωρίς να κάνουμε κάτι περισσότερο. Είναι σημαντικό αυτό και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και με πολλούς άλλους. Θα λοιπόν να σταθώ σε δύο φακέλους ε, και να μου εξηγήσετε γιατί ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αναλάβει δράση. Πρώτον είναι το ζήτημα των φορολογικών παραδείσων και της φοροαποφυγής ε, και γιατί δεν έχετε αναλάβει κάποια δράση έτσι ώστε οι χώρες αυτές που επιτρέπουν τέτοια καθεστώτα να τεθούν πρώτων ευθυνών τους και να μην σταπάψει αυτή η πρακτική. Περιμένουμε κάποια στιγμή να εκφραστεί η θέση της Επιτροπής ε, και να γίνει μια ε, μελέτη των, ε, του αντικτύπου. Αλλά εδώ πρέπει να σκεφτούμε τι θέτουμε στη ζυγαριά. Οι πολίτες απαιτούν φορολογική δικαιοσύνη. Θα το βάλουμε αυτό στο ζύγι με τις ανάγκες των επιχειρήσεων για φορολογική ευηλεξία. Το δεύτερο θέμα είναι το ζήτημα της ε, επισήμανσης της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων των μη αγροτικών ε, προϊόντων βιοτεχνίας. Με γνωμοδότηση ιδίας πρωτοβουλίας ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νομοθετική πρόταση. Εδώ έχουν γίνει πολλές μελέτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει λευκή βίβλο, υπάρχει μελέτη του 2013, υπάρχει πράσινη βίβλο, υπάρχει διαβούλευση με μικρομεσαίε επιχειρήσει και κράτη κτλ. κτλ. Πώς δίνουμε συνέχεια σε όλα αυτά. Η απάντηση της Επιτροπής όταν ερωτήθηκε ήταν χρειαζόμαστε να κάνουμε και άλλε μελέτε Να μελετήσουμε τον αντίκτυπο που θα έχει μια πιθανή υιοθέτηση νομοθεσία πώς μπορούμε να τα συμβιβάσουμε αυτά με τους στόχους που εκθέσατε ως στόχους της Επιτροπής για το ευνομοθετή. Ευχαριστώ κυρία Κάφμαν. Μια σύντομη παρατήρηση και μια σύντομη ερώτηση. Μια παρατήρηση για την διοργανική συμφωνία. Πρέπει να σας πω ότι ε, το αποτέλεσμα με ικανοποιεί, το συζητήσαμε και εδώ στο Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, μελέτες επιπτώσεων. Γιατί γνωρίζετε ότι εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε μια διαφορετική αντίληψη ε, για το αν χρειαζόμασταν ένα εξωθεσμικό, ε, μια εξωθεσμική επιτροπή για να ελέγχει το θέμα αυτό. Πάντως κύριε Τίμερμανς, αν θεωρεί ότι αυτό είναι σωστό, δηλαδή αν η πρόταση ε, της Κομισιόν περιγράφει ένα άλογο και ο νομοθέτης τελικά αποφασίσει ότι χρειάζεται καμήλα, τότε έχει το δικαίωμα να το κάνει. Ε, και μιας και μιλήσαμε για τη συμμετοχή των πολιτών, ενδεχομένως θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για το σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εντός της Κομισιόν διότι υπήρχε και μια έκθεση για την πρωτοβουλία πολιτών και την αναθεώρηση της, ε, του σχετικού ε, κανονισμού. Έχετε προχωρήσει ε, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομε απαντήσει. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κώστα ε, που μα παρατήρησε ότι έχει αυξηθεί η διαφάνεια, έχει βελτιωθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις ε, για διεθνείς συμφωνίες ε, όπως η TTIP. Υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν κάποια όρια γιατί το να αποκαλυφθούν, να δημοσιοποιηθούν κάποια στοιχεία αποδυναμώνει τις διαπραγματεύσεις, τις διαπραγματευτικά μας χαρτιά, γιατί η άλλη πλευρά δεν θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία. Επίσης, στοιχεία τα οποία περιέρχονται στους βουλευτές ε, αν δημοσιοποιηθούν, αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις για ε, να αποκτήσουν κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα ή όφελος. Επομένως, χρειάζεται ε, ένα όριο, ιδίως όσον, όσον αφορά εμπορικής, εμπορικές ε, διαπραγματεύσεις συγκρίνοντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με άλλου διακυβερνητικού οργανισμού ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο άλλο του μεγέθου του, του είδου του οργανισμού που να είναι τόσο διαφανή σε τέτοιε διαπραγματεύσει. Ε, εν τέλει, πάντα θα πρέπει να επιλέγουμε ε, ποια στοιχεία μπορούν να δημοσιοποιηθούν πλήρω, ποια στοιχεία μπορούμε να τα μοιραστούμε με του ευρωβουλευτέ, αλλά ε, στη βάση της εμπιστευτικότητας για να προστατεύσουμε τελικά και τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί έχω εμπειρία από διεθνείς διαπραγματεύσεις, από διαπραγματεύσεις σε διεθνή φόρα, γνωρίζω ότι είναι αποδλήτως αδύνατο να επιτύχει κανείς ένα καλό αποτέλεσμα, ένα ε, αποτέλεσμα ωφέλιμο για, τον, ε, για την πλευρά του, εάν μόνο η δική του πλευρά δημοσιοποιεί στοιχεία, ενώ η πλευρά που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του τραπεζιού λειτουργεί με πλήρη μυστικότητα. Επομένως, κατά περίπτωση κρίνουμε. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της διοικητικής διαδικασίας, ε, εγώ το προσεγγίζω με ανοιχτό πνεύμα, ε, απλώς θέλω να πιστώ ότι εδώ δεν πρόκειται για μία λύση που ψάχνει να βρει πρόβλημα. Θέλω να με πείσετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουμε. Ε, και ότι επίσης ο τρόπος με τον οποίο προτείνεται να το λύσουμε είναι ο ενδεδειγμένος, ότι δεν θα μπορούσε να λυθεί πιο απλά ε, ή με άλλον τρόπο. Με άλλα λόγια σας λέω ότι είμαι ανοιχτό ε, να το συζητήσουμε για το θέμα αυτό χωρίς δογματισμούς. Τώρα, όσον αφορά την αξιολόγηση αντικτύπου. Η αξιολόγηση αντικτύπου δεν είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε αντί των πολιτικών επιλογών. Η αξιολόγηση αντικτύπου είναι ένα τεχνικό ε, έγγραφο, μια μελέτη για να βοηθήσει τους πολιτικούς να λάβουν τις αποφάσεις τους. Όμως ε, συχνά γνωρίζετε ότι το ζήτημα δεν είναι αν ο νομοθέτης επέλεξε άλογο ή Καμίλα. Αυτό που συχνά συμβαίνει είναι ότι εξαιτία των συμβιβασμών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο και των συμβιβασμών με τα 28 κράτη-μέλη, καταλήγουμε να διαλέγουμε Καμίλα ενώ δεν θέλαμε Καμίλα Και δεν χρειαζόμαστε καμήλα. Πολλέ φορέ μα ενδιαφέρει πιο πολύ να επιτύχουμε έναν κάποιο συμβιβασμό παρά το ίδιο το περιεχόμενο του συμβιβασμού. Και αυτοί που κυρίω πλήττονται από αυτή την πρακτική είναι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, είναι οι πολίτε. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά εάν τελικά παραγνωρίζονται, παραμερίζονται ε, τα αναφερόμενα σε μια αξιολόγηση αντικτύπου επειδή αυτό θέλετε να κάνετε, εντάξει. Αλλά να σα δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταλήξει σε μια αξιολόγηση αντικτύπου η οποία λέει ότι μια συγκεκριμένο μέτρο θα οδηγήσει σε κόστο και διαχειριστικό άχθο και τελικά έρθει το Γερμανικό Κοινοβούλιο και επιβάλλει στη Γερμανική κυβέρνηση να περάσει αυτό το μέτρο για πολιτικού λόγου, ε, απλώ να ξέρουμε τι αποφασίσαμε. Αυτό ω απάντηση στην κυρία Γοζιέ για τα δύο ζητήματα ε, που μου ανέφερε για τι αξιολογήσει αντικτύπου. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της ε, Πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών, το ECI, ε, δεν είμαι ακόμα έτοιμο να σα απαντήσω, το εξετάζουμε Ελπίζω να είμαστε σε θέση να σα δώσουμε πολύτερε πληροφορίε στο μέλλον. Ζητώ συγγνώμη που απάντησα έτσι τηλεγραφικά στο τέλο, αλλά πρέπει να φύγω. Ε, έχω ήδη καθυστερήσει. Ο πρόεδρο, ε, σα ευχαριστούμε. Ακούσατε τα θέματα και τι ερωτήσει που σα έθεσαν τα μέλη του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε. Thank you very <laughs> now. Yes, we can do it Okay, uh, before... Λοιπόν, πριν ε, περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, δηλαδή την ανταλλαγή απόψεων με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, την κυρία Ωραϊλή, ε, να σας ενημερώσω για δύο αποφάσεις των ε, συντονιστών. Καταρχάς, η κυρία Χάουταλα είναι η συγκήτρια για την άρση της ασυλίας του Ροζάριο Κροτσέτο και επίσης κύριος Χρυσόγονος είναι υπεύθυνο ε, για την έκθεση, για την αποζημίωση αστικής ευθύνης, ε, για τις ε, παράκτιες διαδικασίες εξόρυξης φυσικού αερίου. Αυτές είναι οι αποφάσεις των συντονιστών. Uh, several seconds before the European Ombudsman enters into the... Λοιπόν, ε, δεν έχει έρθει ακόμα η κυρία Ράιλι, από ότι αφού μείνει εδώ απ' έξω. So shy, omitted. Dear colleagues, we can continue. Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε. Να καλωσορίσουμε May I welcome, uh, Mrs. την κυρία Έμιλι Οράιλι, Ευρωπαία Διαμεσολαβητή Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Να σας ευχαριστήσω κύριε Ράιλι που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για μια ανταλλαγή απόψεων για μια διαδικασία έρευνας που ξεκινήσατε τον Ιούλιο του 2015 και ενδιαφέρει ιδιαίτερο στην Επιτροπή μας. Δεδομένου ότι είμαστε και η αρμόδια Επιτροπή για τη διοργάνωση και ε, το ε, καταστατικό του ε, δικαστηρίου. Ξέρετε ότι είμαστε υπεύθυνοι για το άρθρο 255, τον ορισμό δηλαδή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το τμήμα του ε, Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συγκεκριμένο τμήμα της έρευνας που μας απασχολεί αφορά την άρνηση του Συμβουλίου να δημοσιεύσει τις γνωμοδοτήσεις του πάνελ για τον διορισμό, για το δικαστήριο και για το γενικό δικαστήριο. Αλλά ε, έχω την εντύπωση ότι το θέμα αυτό ε, απασχολεί και γενικότερα και είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητο πλέον ε, το θέμα της διαφάνειας ε, των θεσμικών οργάνων. Θα θέλαμε λοιπόν, πέραν των εξηγήσεών σας για την έρευνα, για τις ε, γνωμοδοτήσεις, ε, για τις ενστάσεις για τους διορισμούς. Θα θέλαμε να μας πείτε και την άποψή σας ε, για το πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη η διαφάνεια και τι ρόλο μπορείτε να διαδραματίσετε εσείς επί του ζητήματος. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε για παράδειγμα σε ποιο βαθμό εσείς σκοπεύετε να κάνετε ανοιχτές διαδικασίες πρόσληψης. Και θα ήθελα τώρα να σας δώσω το λόγο χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Παρακαλώ κύριε Ωράιλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για να έρθω να μιλήσω εδώ σήμερα. Όπως σας έχω πει επανειλημμένως, η σχέση μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ζωτική σημασία και επομένω καλωσορίζω αυτή την πρώτη ευκαιρία να απευθύνω το λόγο εδώ στην Επιτροπή σα. Η αποστολή μου είναι να υπηρετώ την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής ε, ηθικής, διάφανης ε, διοίκησης που λογοδοτεί. Και όλα αυτά σχετίζονται με τη διαφάνεια. Μέσω της διαφάνειας η ευρωπαϊκή διοίκηση μπορεί να είναι υπόλογη προς τους πολίτες που εξυπηρετεί και να αποδείξει στους πολίτες ότι είναι αποτελεσματική και δεοντολογική ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά τους έργανα είναι πάρα πολύ σημαντικά ώστε να έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται την εμπιστοσύνη των πολιτών της, ιδίως σε χαλεπούς καιρούς όπου αντιμετωπίζουμε εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις. Γι' αυτό λοιπόν μετά από την πρόσκλησή σας Σήμερα θα σας πω κάποιες λεπτομέρειες για την έρευνά μου μέχρι τούδε για μια πολύ συγκεκριμένη υπόθεση και θα ακούσω και τις σκέψεις και τις ε, παρατηρήσεις σας για το θέμα. Ε, ξεκίνησε από μια καταγγελία από μια μη κυβερνητική οργάνωση στην ε, Ισπανία την Άξες μη κυβερνητική οργάνωση και ένα μια συνεργασία μεταξύ ε, της νομικής σχολής του Πανεπιστήμιου της Νέας Υόρκης και τη, κάποια σχολή στο Παρίσι. Η συνεργασία αυτή έχει γίνει βάση του άρθρου 225. Ε, είναι ένα πάνελ ε, το οποίο συστήνεται για να γνωμοδοτεί για τους ε, δικαστές και το Γενικό Ισογελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου πριν γίνει ο διορισμός ή ο επαναδιορισμός. Στην έκθεση δραστηριοτήτων δηλώνεται ότι μεταξύ του 2010 και του 2013 το 22% των γνωμοδοτήσεών τους ήταν αρνητικές. Πρέπει να πω τώρα ότι μέχρι σήμερα κάθε γνωμοδότηση, είτε θετική είτε αρνητική, έχει δεχτεί από το Συμβούλιο, κάτι το οποίο επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι το πάνελ και τι επιρροή έχει. Το πάνελ αυτό των 7 επιλέγεται από το Συμβούλιο, από πρώην μέλη του ε, Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, μελών των Εθνικών Δικαστηρίων και εισαγγελέων και ε, κάποιοι εξ αυτών, όπως είπατε, ε, προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο παρέχει τη γραμματεία για το πάνελ. Αυτή τη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να έχει πρόσβαση στις γνωμοδοτήσεις, αλλά το ε, Συμβούλιο αρνείται να δώσει τις ε, ε, γνωμοδοτήσεις. Βάσει τη τρίτη έκθεση δραστηριοτήτων, η γνωμοδότηση συντάσσεται ω εξή. Καταρχά, αναφέρονται τα διάφορα στάδια τη εξέταση. Οι γνωμοδοτήσεις στη συνέχεια αναφέρουν τους λόγους που υποστηρίζουν τις απόψεις του πάνελ, είτε είναι θετικές είτε αρνητικέ, σε σχέση με τις νομικές δεξιότητες, την επαγγελματική εμπειρία, την ικανότητα εκτέλεση των καθηκόντων ενό δικαστή με αμεροληψία και ανεξαρτησία, γνώση ξένων γλωσσών και δυνατότητα εργασίας σε ε, διεθνές περιβάλλον. Το πάνελ πιστεύει ότι οι θέσεις ε, του ε, πάνελ για τις ε, ικανότητες του κάθε υποψηφίου δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δεδομένων, για, την, το αμερόληπτο της διαδικασίας και για διάφορους άλλους λόγους. Αλλά φάνηκε να δέχεται ότι τα πρακτικά καλύπτονται βάσει του κανονισμού 1049 για την πρόσβαση στα έγγραφα. Το πρώτο θέμα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσω εδώ, σε αυτή την καταγγελία, είναι ότι το Συμβούλιο δεν θεωρεί ότι ο κανονισμός 1049, ο κανονισμός δηλαδή για τη δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα, ισχύει για τις γνωμοδοτήσεις του πάνελ. Το πάνελ θεωρήθηκε ότι είναι ένας φορέας ο οποίος συνδέεται με το Συμβούλιο και είναι υπόλογο μόνο προς τα κράτη-μέλη. Εγώ θεωρώ ότι είναι προβληματική αυτή η στάση για διάφορους λόγους. Ο κανονισμός 1049 θέλει να παρέχει την πλήρη δυνατότητα στο μέτρο του δυνατού για πρόσβαση σε έγγραφα. Προφανώς υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά οι εξαιρέσεις πρέπει να ερμηνεύονται με τη στενή του έννοια. Ο κανονισμός 1049 δεν ισχύει. Ε, εάν δεν ισχύει λοιπόν για τα ε, μέλη, για τις νομοδοτήσεις του πάνελ, τι ακριβώς πρέπει να ισχύει και για ποιο λόγο. Η άποψή μου ε, είναι ότι ο 1049 ισχύει για την περίπτωση του πάνελ το Συμβούλιο ε, ενημέρωσε ότι βάσει μιας νέας απόφασης πολιτικής το 1049 ισχύει πλέον για πρόσβαση στα έγγραφα τα οποία διαθέτει η Γενική Γραμματεία όσον αφορά ε, την εκτέλεση υποστηρικτικών καθηκόντων για διάφορες ομάδες όπως για παράδειγμα το συγκεκριμένο πάνελ. Θα ήθελα λοιπόν εδώ επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για την επικοδομητική του απάντηση σε αυτή την πτυχή της ερευνάς μου που οδήγησε σε αυτή την ε, αλλαγή. Επειδή όμω η εσωτερική διαδικασία του Συμβουλίου για τη δημόσια πρόσβαση και τα σχετικά αιτήματα δεν είναι η ίδια με τη διαδικασία που αφορά τις ερωτήσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να απαντήσει όσον αφορά τα αιτήματα για πρόσβαση βάση του 1049 στα πλαίσια της ερευνάς μου. Γι' αυτό ακριβώς, ε, προκειμένου το αίτημα της πρόσβαση να αντιμετωπιστεί βάσει του 1049, οι καταγγέλλοντε θα πρέπει να κάνουν ένα νέο αίτημα πρόσβαση προς το Συμβούλιο αν το επιθυμούν. Εάν δεν δοθεί δημόσια πρόσβαση μετά το νέο αίτημα, θα είμαι σε θέση να ελέγξω ε, αναλυτικά την, το αιτιολογικό του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι η απάντηση του Συμβουλίου προς τους καταγγέλλοντες, παρά το γεγονός ότι δεν βασιζόταν πλήρως στο 1049, υποδηλώνει ότι μπορεί να αρνηθούν να απαντήσουν και σε νέο αίτημα πρόσβασης. Ε, αναφέρονται ανησυχίες για την ε, ε, προστασία δεδομένων και την έκδοση γνωμοδοτήσεών τους. Λέγεται ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις γνωμοδοτήσεις του πάνελ περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της πρόσβασης του 1049 και πρόσβαση των εγγράφων και του κανονισμού 45 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να γίνει μια δοκιμή ισορροπίας λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο δημόσιο συμφόρον και τη διάκριση μεταξύ της έκδοσης αρνητικών γνωμοδοτήσεων και της έκδοσης θετικών γνωμοδοτήσεων. Όλα αυτά είναι θέματα για τα οποία βέβαια δεν μπορώ ακόμα να λάβω θέση. Θα πρέπει να περιμένω ε, το μελλοντικό αίτημα για το ε, ε, δημοσιοποίηση των πληροφορών βάσης του 1049 και σχετική ένσταση και όλα αυτά θα μπορέσω ίσως να τα ξανασυζητήσω μαζί σας εάν οι καταγγέλλοντες κάνουν νέα καταγγελία βάση του 1049 και φτάσει και πάλι στο γραφείο μου ως επίσημη καταγγελία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. Θέλει κάποιο να λάβει τον λόγο, η κυρία Σάιντερ. Κυρία Ρέιντερ; Ευχαριστώ κυρία Διαμεσολαβήτρα που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Νομίζω αυτό το τελευταίο ζήτημα που θέσατε σχετικά με τη διάκριση των θετικών και αρνητικών γνωμοδοτήσεων είναι πολύ σημαντικό. Κατανοώ ότι μια θετική γνωμοδότηση σημαίνει ότι κάποιος ε, θα, μπορεί να ε, διορίζεται. Και σε αυτή την περίπτωση είναι λογικό. Ε, το κοινό, οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν αν η γνωμοδότηση συνάδει με τη συγκεκριμένη απόφαση. Μπορείτε λοιπόν να μας εξηγήσετε σε ποιο βαθμό τα αιτήματα αυτά προς το Συμβούλιο καλύπτονταν ή σε ποιο βαθμό ε, υπήρχαν αρνητικές γνωμοδοτήσεις. Νομίζω ότι ο καταγγέλων ήθελε ε, ε, πρόσβαση σε όλες τις γνωμοδοτήσεις και εξήγησαν τους, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους θεωρούσε ότι θα πρέπει να δημοσιεύονται γνωμοδοτήσεις για λόγους διαφάνειας, ενημέρωση του κοινού και τα λοιπά. Αν το Συμβούλιο αρνηθεί και επανέλθει η υπόθεση σε μένα, το Συμβούλιο λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να δημοσιευθούν πληροφορίες και αν στη συγκεκριμένη περίπτωση ο καταγγέλων επιμείνει όσον αφορά την αξία δημοσίευσης θετικών και αρνητικών γνωμοδοτήσεων θα πρέπει το Συμβούλιο να τεκμηριώσει τη θέση του. Αλλά όπως σας είπα δεν μπορώ να αποφανθώ έως ότου ακούσω ε, όλους τους πιθανούς λόγους. Αυτή τη στιγμή ε, αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι δεν θα ήταν μάλλον ε, κακό να δοθούν στη δημοσιότητα οι θετικές γνωμοδοτήσεις. Με τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο, γιατί ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βλάψει τις προοπτικές καριέρας ενός ανθρώπου στην χώρα του. Όταν δηλαδή... Ε, από την άλλη πλευρά είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το Συμβούλιο Επιλογής ε, θα πρέπει να μπορεί και το ίδιο να υπερασπιστεί τη θέση του και να ε, επιχειρηματολογήσει γιατί οι αποφάσεις που παίρνει είναι ε, τεκμηριωμένες. Φυσικά θα έχετε διαβάσει και τη σχετική έκθεση και προκύπτει ότι η δουλειά που κάνει το συγκεκριμένο Συμβούλιο είναι πάρα πολύ διεξοδική. Σε κάθε περίπτωση, ε, αν το Συμβούλιο αρνηθεί, θα έχω και εγώ την ευκαιρία να ε, έρθω σε επαφή και να διαβάσω την δική του λογική, το δικό του σκεπτικό, γιατί δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες. Η κυρία Χάουτελα, ευχαριστώ και σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Έχω μια γνώμη, μια άποψη που θα ήθελα να σας εκφράσω και δύο ερωτήματα. Όταν ε, ήμουν στην κυβέρνηση της χώρας μου, υπεύθυνοι για την επιλογή ενός γενικού γραμματέα μεταξύ πολλών υποψηφίων, ήμασταν υποχρεωμένοι να δημοσιεύσουμε ένα πίνακα με συγκριτικά στοιχεία των υποψηφίων βάσει του οποίου τελικά είχαμε καταλήξει στην απόφαση διορισμού μας. Και αυτό φυσικά έδινε, ε, αποκάλυπτε και πολλά θέματα, πολλές πλευρές της ε, γνώμης που είχαν σχηματίσει ε, τα μέλη της Επιτροπής για τον εκάστοτε υποψήφιο. Και δεν ξέρω αν ήταν 100% θετικό ε, η διαδικασία, ήταν 100% ε, θετική η διαδικασία αυτή. Μπορείτε να αναλύσετε όσον αφορά την αυτογλωκοκρισία έχετε δίκιο σε αυτά που είπατε και κάτι ακόμη ε, πριν από λίγη ώρα είχαμε συζήτηση με τον κύριο Τίμερμανς για ορισμένα συζητήματα διαφάνειας και τέθηκε το θέμα ότι ε, υπάρχει μια ισορροπία που πρέπει να επιτυχάνεται μεταξύ αποτελεσματικότητας και διαφάνειας. Για παράδειγμα όσον αφορά την δημοσίευση εγγράφων που χρησιμοποιούνται στον τριμερή διάλογο. Ξέρω ότι δεν συζητούμε σήμερα ακριβώς αυτό, αλλά μήπως θα μπορούσατε εσείς να μας ε, πείτε δύο λόγια για το πώς χειρίζεστε αυτό το θέμα, το θέμα της διαφάνειας στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο τρόπος που το πάνελ το κάνει δεν είναι ότι συγκρίνει ε, με μονομερμένες υποψηφιότητες, αλλά εξετάζει την κάθε υποψηφιότητα ε, αυτόνομα. Φυσικά ε, εξετάζονται ε, και οι άνθρωποι που πρόκειται να παραταθεί η θητεία τους. Όσον αφορά αυτό το, αυτή την αυτολογοκρισία που είπατε, φυσικά ορισμένες φορές στη διαδικασία κάποιου ελέγχου αυτό είναι απαραίτητο και σε αυτό αναφερόμουν. Όσον αφορά αυτό που είπατε για τους τριμερείς διαλόγους, όπως γνωρίζετε, ε, βρίσκεται σε εξέλιξη μια έρευνα από πλευράς μας για τη διαφάνεια στους τριμερείς διαλόγους και αυτή ξεκίνησε λόγω ανησυχιών που εκφράστηκαν ε, ε γι' αυτό που κάποιοι θεωρούν ότι αποτελεί έλλειψη διαφάνειας είναι πράγματι πολύ αποτελεσματική διαδικασία η τριμερής διάλογη αν κρίνει κανείς από τον όγκο των νομοθεσιών που εγκρίνονται εκεί και στην ε, ακαδημαϊκή βιβλιογραφία ε, η οι τριμερής ε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξισορρόπησης αποτελεσματικότητας και διαφάνειας. Πολλές φορές συνάδελφοί μου έχουν παρακολουθήσει τους τριμερείς διαλόγους για να διαπιστώσουν τι ακριβώς τελικά δημοσιεύεται και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε στενότερα το ζήτημα των δημοσίων διαβουλεύσεων. Άρα, όπως είπε μάλλον και ο κύριος Τίμερ μας, ε, είναι πραγματικά ένα θέμα ε, πού ακριβώς θα θέσει κανείς τον πύχη και πού ακριβώς θα θέσει την, την κόκκινη γραμμή. Ε, εγώ ήμουν επίτροπος στην Ιρλανδία και όποτε πήγαινα στο Εθνικό Κοινοβούλιο έλεγα ότι η διαφάνεια, στόχος της διαφάνειας δεν είναι να ε, προκαλέσει προβλήματα. Και αυτό όπως και το ζήτημα της δημοσίευσης των γνωμοδοτήσεων, θα πρέπει να ε, ε, το προσεγγίζει κανείς πάντοτε υπό αυτό το πρίσμα. Ε, το αν δηλαδή είναι θετικό να δημοσιευθούν οι θετικές και αρνητικές γνωμοδοτήσεις και ενδεχομένως κάτι τέτοιο θα μπορούσε ίσως να βλάψει την ίδια τη διαδικασία ή θα μπορούσε να αποτρέψει ανθρώπους από το να θέτουν υποψηφιότητα. Άρα αυτό συνολικά δεν θα κρινόταν ε, ως κάτι το θετικό. Πάντως, εκτός από τη σημασία των δικαστικών αποφάσεων, το ζητούμενο για το πάνελ ήταν ότι, στις, ε, ότι σε διάφορες χώρες ακολουθούνται διάφορες διαδικασίες για τον διορισμό των δικαστών. Σε κάποιες χώρες είναι εντελώς διαφανής η διαδικασία, σε άλλες λιγότερο διαφανής. Το πάνελ αυτό που προσπάθησε να κάνει είναι να αφαιρέσει όλους αυτούς τους παράγοντες και να εξετάσει τις υποψηφιότητες και τους διορισμούς στη βάση των προσόντων του κάθε υποψηφίου και από αυτή την άποψη ε, θεωρούμε, θεωρώ ότι ήταν μια θετική διαδικασία. Η κυρία Ντελβό, σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να θέσω κάποιο ερώτημα. Μια και όμως ρωτήσατε ποια είναι η άποψή μας, θέλω να εκφράσω κι εγώ τη δική μου. Αντιλαμβάνομαι όλα αυτά τα αιτήματα, όλες αυτές τις εκκλήσεις για διαφάνεια και τις υποστηρίζω. Τις υποστηρίζω για θέματα όπως η TTIP κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε για τα προσόντα ατόμων. Και εδώ πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι αν θέλετε. Και γι' αυτό ε, χαίρομαι που είπατε ότι η διαφάνεια δεν θα πρέπει να προκαλεί βλάβη. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη δημοσιοποίηση ε, νομοδοτήσεων, πορισμάτων που τελικά αφορούν τα προσόντα κάποιου ανθρώπου. Μπορώ να αντιληφθώ γιατί να δημοσιοποιηθεί μια θετική γνωμοδότηση αλλά σε καμία περίπτωση μια αρνητική γνωμοδότηση, η οποία μάλιστα θα μπορούσε να βλάψει και την επαγγελματική σταδιαδρομία αργότερα του ιδίου προσώπου. Ε, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Φαντάζομαι ότι δεν θα, έχουν, δεν θα επιθυμούσαν και ξαφνικά θα δημοσιοποιηθούν και όλα τα σε δυναμίες τους όλα τα αρνητικά του στοιχεία. Επομένω, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τους περιορισμούς, με την στάθμιση ε, του, που θα μα οδηγήσει στο να αποφασίσουμε αν θα δημοσιοποιούνται αυτά τα στοιχεία. Ο κύριος Λεπδετό. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το ζήτημα που συζητάμε σήμερα έχει τεράστια σημασία γιατί η διαφάνεια έχει τεράστια σημασία για τις δημοκρατικούς θεσμούς. Και ανησυχώ με αυτά που ακούω για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Λίγο πριν ο, ο αντιπρόεδρος Τίμερμαντς προσπάθησε να μας καθησυχάσει αλλά στην πραγματικότητα καταλήξαμε στο να καταρτήσουμε ένα κατάλογο με όλους τους τομείς τους οποίους δεν υπάρχει διαφάνεια. Η TTIP, οι άλλες διεθνείς διαπραγματεύσεις για τις υπηρεσίες, και άλλα θέματα στα οποία η διαφάνεια σταματάει με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Και εδώ, στο αυτό το σημείο της μερικής διάταξης, διακυπιστώνουμε ότι το Συμβούλιο προσπαθεί με ερμηνείες των κανονισμών διασταλτικές να περιορίσει την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία, σε ορισμένα, να, την διαφάνεια σε αυτά τα στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και με την περίπτωση όπου φάκελοι ε, δεν ε, φτάνουν στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα και διαπιστώνουμε ότι ούτε καν και οι τριμερείς διάλογοι, στους οποίους εκπροσωπούνται και τα τρία θεσμικά όργανα, δεν είναι απολύτως διαφανείς. Σέβομαι τον θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, εσάς κύριε Ράιλι, γιατί εσείς πραγματικά συνεισφέρετε στην διαφάνεια. Ωραία. Αυτές ήταν τοποθετήσεις, θετικές τοποθετήσεις και όχι ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Ράντα, θέλετε το λόγο πάλι. Ναι. Με την άδειά σας και αν έχουμε το χρόνο. Μιας και έχει τεθεί το ζήτημα του εάν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται οι αρνητικές γνωμοδοτοδιστήσεις εγώ δεν έχω κατασταλάξει ακόμα. Γιατί θα μπορούσε κανείς να πει ότι συγκρίνοντας μια θετική γνωμοδότηση και μια αρνητική γνωμοδότηση μπορούμε να εξάγουμε και από αυτό συμπεράσματα. Θα ήθελα κάποια περισσότερα στοιχεία. Τι συμβαίνει συνήθω, Συμβαίνει συχνά να έχουμε αρνητικέ γνωμοδοτήσει, είναι μάλλον η εξαίρεξη. Αυτό επίση νομίζω έχει σημασία για να σκεφτούμε εάν πραγματικά το δημόσιο συμφέρον εδώ υπερισχύει. Δηλαδή, εάν πολύ σπάνια τυχαίνει κάποιος υποψήφιος να απορριφθεί και να έχει μια αρνητική γνωμοδότηση ε, και αυτό επειδή πολύ συχνά οι υποψήφοι ε, έχουν πολύ ψηλό επίπεδο προσόντων, ε, τότε θα ήταν λογικό να να, να περιμένουμε, να, να υποθέσουμε ότι η δημοσιοποίηση της αρνητικής γνωμοδότησης θα έχει αρνητικά ε, αποτελέσματα. Ανάμεσα στο 2010 και στο 2013, το 22% των γνωμοδοτήσεων ήταν αρνητικές, ενημερώνει η κυρία Οράιλη. Συνολικά, το 22% ήταν αρνητικές. Οι υπόλοιπες ήταν ε, και στην περίπτωση μάλλον τη ανανέωση θητεία ήταν πάντα θετικέ, ήταν όλε θετικέ. Επομένω, δεν ε, εγκρίνονται όλε οι υποψηφιότητε ε, αυθορή αλλά ε, σε μεγάλο βαθμό εγκρίνονται. Ο πρόεδρο φαίνεται ότι έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση και για αυτό το θέμα τη ημερήσια Έταξη. Ευχαριστούμε την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια για αυτή την ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. στο πλαίσιο είναι αναρμοδιοτήτων τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου για την ε, ορισμό των ε, δικαστών του, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σα ευχαριστούμε για την παρουσία σα εδώ. and we can continue by Okay, uh, let us continue by point number... Ωραία. Να συνεχίσουμε με το σημείο 13. και βρίσκεται εδώ ο εισηγητής. Μιλούμε για τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και θα εξετάσουμε το έγγραφο εργασίας. Δίνω το λόγο στον εισηγητή. Ε, muchas gracias, señor presidente. Distinguidos κολέγας, En este segundo documento de αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για την δεύτερη, για το δεύτερο έγγραφο εργασίας που υποβάλλω σε εσά προς εξέταση και μπορώ να σας πω ότι μέχρι στιγμής το έργο μας για αυτήν την πρόταση ε, βαίνει καλός ε, για τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύσεις Θα τα πω λίγο τηλεγραφικά. Μιλήσαμε ε, έχουμε, ε, στις 19 Απριλίου 2014 υπευλήθη η πρόταση. Λίγο αργότερα εντός της ίδιας χρονιάς ορίστηκε εισηγητής ε, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για να παρακολουθεί το θέμα. Τον Δεκέμβριο του 2014 σε αυτήν την Επιτροπή έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και έκτοτε φάνηκε ότι υπήρχε πολύ ισχυρή διαφωνία ευρωβουλευτών με αυτήν την πρόταση και την βιωσιμότητα της. Παρ' όλα αυτά συνεχίσαμε να ε, εργαζόμαστε επί της πρότασης αυτή για να παρακολουθούμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Το 2015 ε, υπευλήθη και ένα έγγραφο εργασίας το οποίο ήρθε να ενισχύσει τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί στο, στην Επιτροπή μας. Πάρα, πολύ, ε, πάρα πολλές οργανώσεις, συνδικάτα, καθηγητές πανεπιστημίου ε, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για αυτήν την πρόταση και εμείς έχουμε διοργανώσει πολλές συναντήσεις μεταξύ των συντονιστών και έχουμε ειλικρινεί ε, συζητήσεις διεξαγάγει για να καθορίσουμε ποιος θα ήταν ο τρόπος που θα χειριζόμασταν το ζήτημα αυτό. Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς υιοθέτησε μια ε, προσέγγιση και εγώ προσωπικά ε, συμφωνώ ιδιαίτερος με αυτήν την στάση της συγκεκριμένης Επιτροπής. Δεν ε, ήθελα να σταματήσω γιατί υπήρχαν αρκετοί ε, εισηγητές και συνάδελφοι που μου ζήτησαν να συνεχίσω. Αυτή είναι η τελευταία παρουσίαση και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουμε τις διάφορες διαδικασίες. Ε, να καλέσουμε τους κοιόδης εισηγητές, ε, οι οποίοι βοήθησαν και εδώ, να τους διαβουλευτούμε ώστε να μας δώσουν τα σχόλιά τους και ε, αφού ακούσουμε τα απόψεις τους και γίνει μια σύντομη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και να κλείσει ο κύκλος αυτού του σχεδίου έκθεσης. Προς το καλό ή προς το κακό. Αλλά τέλος πάντων ε, ε, ούτως ή άλλως η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Τώρα επιτρέψτε μου να σας περιγράψω τα ουσιαστικά στοιχεία των αλλαγών που περιλαμβάνει το ε, έγγραφο εργασίας. Όλες οι αλλαγές ε, είναι λόγω των ενστάσεων που εξέφρασαν ε, οι σκιώδεις συζητητές ή των απόψεων που εξέφρασαν όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά είναι τα ουσιαστικά στοιχεία. Αναφέρονται πιο αναλυτικά στο έγγραφο. Θα προσπαθήσω βέβαια να σας τα πω γιατί μπορεί να μην είχατε χρόνο ή θέλετε να επικεντρωθείτε λίγο περισσότερο ε, και να τα ακούσετε. Λοιπόν, καταρχά, ε, ε, θα θέλαμε να περιορίσουμε αυτέ τι μονοπρόσωπε εταιρείε περιορισμένη ευθύνη στι πολύ μικρέ και στι μικρέ επιχειρήσει. Αυτέ που έχουν κάτω από 50 υπαλλήλου και έχουν μικρό κύκλο εργασιών και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε πραγματικά να αποφύγουμε να δημιουργηθούν ε, κάποιες πλασματικές επιχειρήσεις, εικονικές επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα χρήματος. Επίσης θέλουμε να προσδώσουμε μεγάλη αξία στις ε, νεοφυείς επιχειρήσεις, στις start-up, ε, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες επιχειρήσεις καινοτόμε και γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να γίνουν μονοπρόσωπες εταιρείε ε, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο επιχειρηματικής διαδικασίας. Αυτό αναφέρουν τα άρθρα 7, 8 και 9. Το άρθρο 10 περιλαμβάνει μια τροποποίηση από πλευρά τη πρώτης τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου και δίνουμε και ένα βήμα παρατέρω, ώστε ε, κάποιε επιχειρήσει που να θέλουν να λειτουργήσουν ω μονοπρόσωπε εταιρείε περιορισμένη ευθύνη να έχουν συγκεκριμένη έδρα, ώστε να μην γίνεται απάτη έδρα που θα μπορούσε να οδηγήσει και φοροδιαφυγή. Όλα αυτά είναι μια αλλαγή η οποία πραγματικά έπρεπε να γίνει και θέλουμε η σύσταση να γίνεται, της επιχείρησης αυτής να γίνεται διαδικτυακά και ώστε να υπάρχει και ένα ηλεκτρονικό μητρό επιχειρήσεων. Επίσης, σε περίπτωση που υπάρχει υποψία πάτης, ε, θα μπορούμε να ζητούμε φυσική παρουσία του ιδρυτή της επιχείρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13, και επίσης να μπορεί ε, να διαλυθεί η επιχείρηση σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η επιχείρηση δεν, διαρκεί καμία, ε, δεν ασκεί συγγνώμη, καμία επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τη σύσταση μιας ε, ε, επιχείρησης βάσει της πρότασης προτείνουμε ένα ενίο υπόδειγμα καταστατικού. Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 11. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για τα συγκεκριμένα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται και όλα αυτά τα συνδυάζουμε με τις πληροφορίες που θα μπορούν να ζητήσουν τα κράτη-μέλη ε, για το μητρό των επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 13. Ένα άλλο από τα ουσιαστικά στοιχεία είναι να συγχρονίσουμε τη διαδικασία. Εδώ έχουμε το μεταχικό κεφάλαιο στο άρθρο 16. Να μπορεί κάποιο να συστήσει μια εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 1 ευρώ, αλλά να υπάρχουν κάποιε νομικέ υποχρεώσει υποχρεωτικά και ώστε να διασφαλίζεται η αγαστή λειτουργία αυτή τη επιχείρηση. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα μπορούσα να συνεχίσω να σα εκθέτω όλε τι προτάσει μα, αλλά φαντάζομαι ότι είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε αυτό το έγγραφο εργασία και να εξετάσετε ενδελεχέστερα όλε τι πτυχέ που σα ενδιαφέρουν. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τι με ενέπνευσε να κάνω όλε αυτές τις αλλαγές. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου η ανεργία ορισμένες φορές μετατρέπεται σε αυτοαπασχόληση για τους νέους ανθρώπους που δεν ε, ε, προσπαθούν να βρουν μια θέση εργασίας σε ευνοϊκό κλίμα και δεν έχουν εγγυήσεις για έναν αγαστό εργασιακό βίο. Ε, και ε, υπάρχουν πάρα πολλοί εφάνταστοι νέοι που κάνουν ε, κάποια καινοτόμα πράγματα. Θα πρέπει όμως να υπάρχουν κίνητρα για να συστήσει κάποιος μια επιχείρηση και φυσικά στην ψηφιακή εποχή πρέπει να υπάρχουν μέτρα στην νομοθεσία που να επιτρέπουν αυτές τις καινοτομίες. αυτό είναι το πνεύμα που διέπει και την Επιτροπή Γιούγκερ και εμείς ακολουθούμε αυτό το πνεύμα διότι θεωρούμε ότι αυτό μας περιμένει στο μέλλον. Εγώ έκανα ε, την προσπάθεια με ιδιαίτερη ε, αφοσίωση όσο μπορούσα. Δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω γιατί δεν συμμετείχα στις συγκεκριμένες ιδέες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπόρεσα να, να συμφωνήσω επίσης και με τις αμφίσιμες ιδέες του Συμβουλίου γιατί θεωρώ ότι ήταν και λυπής. Και επίσης, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπόρεσα να ακολουθήσω αυστηρά ε, όλες τις συστάσεις των σκιωδών εισηγητών. Και δεν μπόρεσα επίσης να ακολουθήσω και κάποιους συναδέλφους που επειδή ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο ζήτημα έκαναν τις συστάσεις τους. Ευτυχώ όμω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για, διακρίνεται για κάτι, για την διαφάνειά του και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι ε, όλοι μπορούν να ε, μιλήσουν με τον ε, εισηγητή, του λένε αν το θεωρούν κάτι θετικό ή αρνητικό και λόγω των προσωπικών του οικονομικών εμπειριών ή και λόγω των πολιτικών του πεπιθήσεων. Εγώ λοιπόν όπω σα είπα και στην αρχή θέλησα με το έγγραφο αυτό να κάνω μια τροποποίηση και να έχουμε μια ελάχιστη δυνατή συνένεση ώστε να μας οδηγήσει φυσικά σε ένα κείμενο το οποίο βεβαίως και θα έχει και τροπολογίες και θα αλλάξουμε το κείμενο, θα το συμπληρώσουμε, θα το βελτιώσουμε αλλά επιμένω ότι ε, για ε, συγκεκριμένους ιδεολογικούς λόγους ή και για συγκεκριμένους προκαθορισμένους πολιτικούς λόγους ή και μετά από την ανάλυση αυτού του δεύτερου και τελευταίου κειμένου θεωρήσετε ότι δεν μπορείτε να το υποστηρίξετε, πρέπει να λάβουμε μια απόφαση. Υπάρχει προηγούμενο άλλωστε. Ορισμένες φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει και η ε, πραγματικότητα είναι αυτή η οποία επιτάσσει τι πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία του να διαμορφώσουμε μία ε, νομοθεσία επιχειρήσεων ε, μπορεί να μας οδηγήσει και πάλι σε, για πολλωστή φορή, φορά σε ε, αποτυχία. Ε, αποσύρθηκε η πρόταση για την ευρωπαϊκή επιχείρηση, τώρα αλλάζουμε εκ την πρόταση και ίσως θα ε, πρέπει να το συνειδητοποιήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν υπάρχει επαρκή συνένεση, ίσω θα έπρεπε να αλλάξει όλο το επιχειρηματικό σύστημα με μία πρόταση που ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρήσει ότι αξίζει και να ασχοληθούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα σχόλιά σα, ευχαριστώ και για τι απόψει ε, που θα ε, εκφράσετε είτε θετικέ είτε αρνητικέ προ τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Mrs. Regner. Η κυρία Ρέγνερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προτού θέσω ε, το ερώτημα που θέλω και πρωτού κάνω κάποιες παρατηρήσεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την απίστευτα υπομονετική του στάση. Η κατάσταση είναι κάθε παρά εύκολη και απλή. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχουμε ασχοληθεί επιμακρών με το συγκεκριμένο θέμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον εισηγητή, γιατί με πολύ επικοδομητικό τρόπο προσπαθεί πάντοτε να λάβει υπόψη του όλες τις απόψεις που εκφράζονται. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις για το έγγραφο. Και συγκεκριμένα, ε, θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα. Το ζήτημα της ε, επαγγελματικής έδρας. Το ζήτημα με τις εικονικές έδρες και τις εταιρείες σφραγίδες ή γραμματοκιβώτια που χρησιμοποιούν πολύ για λόγους φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής. Δεν ξέρω αν η διατύπωση του άρθρου 10 έχει γίνει κατανοητή από μένα. Εδώ αναφέρεται ότι η, και η κύρια ε, έδρα ε, της εταιρείας συμφωνεί με την πραγματική ε, έδρα της εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υποχρέωση η διοικητική έδρα και η οικονομική έδρα, η έδρα των, της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης να ταυτίζονται. Μου φαίνεται δηλαδή ότι η πρόθεση είναι αυτή με την οποία θα συμφωνούσα και εγώ βεβαίως, αλλά θα ήθελα να ε, μου εξηγήσετε επακριβώς τι ακριβώς σημαίνει η συγκεκριμένη διάταξη και η συγκεκριμένη διατύπωση. Για τα πιο συγκεκριμένα σχόλια που θα ήθελα να κάνω, να πω τα εξή. Πρώτον, για το πεδίο ισχύω, θεωρώ ότι είναι πολύ ικανοποιητικό το γεγονός ότι ε, λόγω και της ανησυχίας που έχουμε ε, ε, εκφράσει. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Είμαι ένα νομικό πρόσωπο και αξιοποιώ αυτό το εργαλείο με τρόπο που δεν εντασσόταν εντός των προθέσεων του νομοθέτη και γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ ε, μιλούμε για επιχειρήσεις που έχουν έως 50 εργαζομένους, υπαλλήλου. Εδώ όμως υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος για όλον τον γεωργικό κλάδο, γιατί πολλές φορές ε, υπάρχουν πολλές ε, μικρές επιχειρήσεις στον συγκεκριμένο τομέα όπου υπάρχει κίνδυνος να συνεχίσουν ε, συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί κύκλοι να χρησιμοποιούν αυτό το, το νομοθέτημα ε, καταχρηστικά. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχει η εταιρεία McDonald's. Θέμα που συζητήσαμε και στο πλαίσιο της Επιτροπής για τις φορολογικές αποφάσεις και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για ε, δομές επιχειρηματικές που ε, λειτουργούν με τη μέθοδο του franchising. Άρα μιλούμε πάντοτε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, τυπικά. Άρα ενδεχομένως και σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να υπάρξει κατάχρηση του νομοθετήματος σε αυτή την περίπτωση. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι το ζήτημα της ε, διαδικτυακής καταχώρησης. Αναφέρεται λοιπόν ότι θα πρέπει ο ιδρυτής μιας επιχείρησης να ε, παρουσιάζεται αυτοπροσώπος στην ε, αρμόδια αρχή, αλλά εδώ υπάρχει το πρόβλημα της εφαρμογής. Υπάρχουν τόσοι πολλοί τομείς που έχουμε ρυθμίσει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου ερχόμαστε εκ των υστέρων και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την εφαρμογή των ε, κανόνων που έχουμε θεσπίσει. Και τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς κομισιών. Ακριβώς επειδή έχει ήδη αφιερωθεί τόσος χρόνος και τόση ενέργεια στο συγκεκριμένο θέμα να στεφθεί κάποια στιγμή με επιτυχία και να καταλήξει κάπου. Ωστόσο, πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι στην ε, σχετική συζήτηση συμμετέχουν ε, κατά πλειοψηφία εκείνοι που είναι υπέρ αυτών των μονοπρόσωπων εταιρεών. Και από αυτή την άποψη εγώ πιστεύω ότι παρά τις εξαιρετικά συμβιβαστικής στάσεις που επέδειξε ο εισηγητής ότι η καλύτερη λύση είναι να απορρίψουμε το, τη συγκεκριμένη ε, πρόταση και να ζητήσουμε να υποβληθούν νέες προτάσεις που θα αφορούν το συγκεκριμένο θέμα της μορφής των ε, εταιριών και της έδρας των εταιριών. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Χάουταλα και σας παρακαλώ να είστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Σας ευχαριστώ. Έχω ασκήσει σφοδρή κριτική στην αρχική πρόταση της Κομισιόν και χαίρομαι που ο εισηγητής έκανε προσπάθειες να ε, διορθωθούν οι κυριότερες ανησυχίες, να αντιμετωπιστούν τα κυριότερα προβλήματα. Ανάμεσα σε αυτά είναι για παράδειγμα οι κεφαλαϊκές απαιτήσει, οι οποίες επιβάλλονταν στις ε, ε, εταιρείε αυτής της φύσεως. Η πρόταση της Επιτροπής στο θέμα αυτό δεν ήταν επαρκής. Επίσης έχουμε ασκήσει κριτική στο ζήτημα το διαχωρισμό των εδρών. Τώρα, είναι προφανές ότι δεν είναι εύκολο, δεν είναι δυνατόν μάλλον, να προταθούν λύσεις οι οποίες να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί για πολλά από τα θέματα στα οποία αναφέρεται αυτή η νομοθετική πρόταση υπάρχει εθνική νομοθεσία πολύ διαφορετική. Επομένω φοβάμαι ότι αυτή η πρόταση τελικά θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο κατακαιρματισμό και πολυπλοκότητα γιατί θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εθνική νομοθεσία. Και τίνω να σκέφτομαι αυτό που είχαμε πει και στην αρχή ότι προτού ε, έχει νόημα να συζητήσουμε για μια τέτοια πρόταση και να είναι μια τέτοια πρόταση χρήσιμη. Πρέπει πρώτα να γίνει μια αναθεώρηση ε, του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου που είναι και το πλαίσιο. Θα το συζητήσω το θέμα αυτό με τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Απασχόλησης που ήταν και η κύρια Επιτροπή που ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό αλλά Συγχαίρω τον συγγητή για τη δουλειά που έκανε, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την πρόταση αυτή της Επιτροπής. Ευχαριστούμε κύριε Ιούδελαντ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να πω προς τον εισηγητή ότι η όποια κριτική ασκούμε στην πρόταση αυτή δεν προπηγάζει από ιδεολογικές διαφορές, αλλά από μια αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων και από ανησυχία. Χαίρομαι που η συγητής μας παρουσιάζει την προσθήκη κάποιων περισσότερων ε, ασφαλιστικών δικλείδων στην στην πρόταση, αλλά δεν αρκούν. Για παράδειγμα, δεν έχουμε εξασφαλίσει ότι αυτή η νομοθετική πρόταση δεν θα μπορούσε να ε, τύχει αντικείμενο εκμετάλλευση ε, για εταιρείε οι οποίε θέλουν να την να, να διαπράξουν ε, απάτη. Διαδικασίες online εγγραφής εταιριών στο Μητρό θα διευκολύνουν τέτοιες παράνομες πρακτικές. Ακόμα και αν δώσουμε στα κράτη-μέλη το δικαίωμα να απαιτούν την φυσική παρουσία του εγγραφόμενου, δεν θα έχουν κανένα τρόπο να το ελέγχουν στην πράξη αυτό. Και αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα όταν ο ετών βρίσκεται στο εξωτερικό. Όπως σας είχα ενημερώσει, την... πρόσφατα η Σουηδική Σουηδικές εταιρείες έστειλαν ε, επιστολή προς τον Σουηδό Υπουργό ε, Δικαιοσύνης με την οποία εκφράζουν μια σειρά ανησυχιών ε, και αντιδρούν στη δημιουργία αυτού του νέου τύπου εταιρείας. Αυτή η απλοποιημένη εταιρική μορφή θα μπορούσε να δημιουργήσει όλο και περισσότερες εταιρείες φαντάσματα ε, και επίσης ε, κλοπή ταυτότητας. δεν θα υπάρχει κάποιο φυσικό πρόσωπο στο οποίο, για παράδειγμα, να επιδίδονται δικαστικές κλήσεις, αποφάσεις που να λογοδοτεί, που να εκπροσωπεί την εταιρεία. Επίσης με τις κεφαλαϊκές απαιτήσει αυξάνεται το ε, ενδεχόμενο ε, απάτης. Ε, αυτή η πρόταση θα διευκολύνει την πιθανότητα διάπραξης τελικά οικονομικών εγκλημάτων. Οι σουηδικές υπηρεσίες, μυστικές υπηρεσίες έχουν επίσης εκφράσει την ανησυχία τους ότι θα μπορούσε αυτή η μορφή εταιρεία να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Θα ήθελα, ε, ακούσει αυτά τα στοιχεία, να έχουμε και την άποψη της Eurojust και της Europol. Έχουν εξετάσει αυτές οι υπηρεσίες ε, την πρόταση για τις μονοπρόσωπες της Επιτροπής από τη δικιά τους σκοπιά θα είχε νομίζω κάποια αξία να γνωρίζουμε και τη δικιά τους άποψη. Ιδιαίτερα σε αυτές τις περιόδους που έχει ε, ενταθεί η τρομοκρατία. Για όλους αυτούς τους λόγους, για όλες αυτές τις ανησυχίες που σας περιέγραψα και εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι σήμερα, ε, ανησυχούν πραγματικά και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω πραγματικά από τον εισηγητή, τον ε, κύριο Καρσία Πασκάλ, Γκράντες Πασκουάρ, να ε, αποτρέψει τη συνέχεια της συζήτηση για αυτή την ε, ε, ε, πρόταση της Επιτροπής. Σε ευχαριστούμε κυρία Γοζιέ. Ευχαριστώ. Υπήρχαν προβλήματα και ανησυχίες από την αρχή που ξεκινήσαμε να εξετάζουμε το κείμενο αυτό και συνεχίζουμε να μην έχουμε λάβει υβρή απαντήσεις. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά του εισηγητή, αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης ερώτηση, ένα θεμελιώδες ερώτημα ε, προς την Επιτροπή, που είναι το εξής. Τι προσπαθούμε να λύσουμε με αυτό το νομοθέτημα. Γιατί χρειάζεται να δημιουργήσουμε αυτή τη νομική μορφή, γιατί χρειάζεται μια μικρή επιχείρηση να δημιουργήσει θηγατρική εταιρεία σε άλλο κράτος μέλος για να δραστηριοποιηθεί διασυνοριακά. Γνωρίζω μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται συνοριακά, δεν βλέπω γιατί τους χρειάζεται μια τέτοια δομή. Ίσως η απλοποίηση των διασυνορικών διαδικασιών να, να, να μπορεί να βοηθήσει τέτοιες επιχειρήσεις. Δεν βλέπω όμως γιατί η δημιουργία αυτής της, ε, μικρο, ε, της μορφής, της μονοπρόσωπης την προτείνει η Επιτροπή, θα μας βοηθήσει. Διαπιστώνουμε μάλιστα ότι οι ίδιες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εναντίον της πρότασης γιατί θεωρούν ε, ότι αυτό το σύστημα θα ανοίξει ακόμα μια, ε, ένα παράθυρο για ε, φορολογική φοροποφυγή και άλλες μορφές οικονομικών εγκλημάτων. Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί τελικά οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν υποστηρίζουν μια πρόταση που υποτίθεται ότι κατατίθεται προ όφελό του. Και το άλλο ερώτημα που ε, ακολουθεί είναι ότι αν δεν βοηθάει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, τελικά ποιον βοηθάει. Χαιρετίζω την προσπάθεια του εισηγητή, ο οποίο έχει προσπαθήσει να βρει απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα ε, και να προσθέσει και άλλες, ε, άλλα στοιχεία που να εξασφαλίζουν τις ανησυχίες που, έχουν εκφράσει, που έχει εκφράσει το Κοινοβούλιο. Αλλά οι ουσιώδεις διατάξεις δεν έχουν τροποποιηθεί. Τώρα, εάν λέμε ότι θα εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο το εθνικό δίκαιο, ότι πολλέ από τι περισσότερε διατάξει τελικά θα παραμένουν στο εθνικό δίκαιο, ε, στην πραγματικότητα τι προσθέτει αυτή η πρόταση και σε τι διαφέρει από την πρόταση για SUP. Σε ορισμένε περιπτώσει μάλιστα δεν είναι ξεκάθαρο ε, ποιο δίκαιο εφαρμόζεται. Το δίκαιο στο οποίο έχει εγγραφεί η μητρική ή στο δίκαιο στο οποίο εφαρμόζεται τη χώρα που έχει εγγραφεί η δικατρική εταιρεία. Είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά ευαίσθητο και αυτό. Επίσης οι μενοπρόσωποι, ε, το, μοναδικό πρόσωπο που εχει εγγραφει η δικατρικη εταιρεια ειναι ενα ζητημα εξαιρετικα ευαισθητο και αυτο επισης οι το μοναδικο προσωπο που ειναι ο εταίρος της ΕΠΕ αυτής εντάξει, εάν πρόκειται για ένα φυσικό πρόσωπο, να το καταλάβω. Αλλά γιατί να μην επιτρέψουμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το εργαλείο αυτό, αν το θεωρούμε καλό, ε, Αντιθέτως προβλέπω ότι στην πραγματικότητα θα, θα, δημιουργηθούν πολλές εταιρείε βιτρίνα. Δεν θα βοηθήσει πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά την φοροαποφυγή. Επομένω, τα προβλήματα που είχαμε εκφράσει στην προηγούμενη πρόταση για το SUP παραμένουν και στην τωρινή πρόταση. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γίνεται πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους προλαλήσαντες ε, για την ε, συνεισφορά τους. Ο εισηγητής ε, προσπαθεί όντως να λάβει υπόψη όλες τις απόψεις. Η συζήτηση όμως αυτή είναι ανούσια. Είναι πολύ δύσκολο να την κατανοήσουμε και ε, γινόμαστε δημαγωγοί, τρομοκρατία για τις μονοπρόσωπες εταιρείε. Όταν συζητούσαμε το PNR και την ανάγκη εισαγωγή ε, του PNR, η αριστερά ήταν ε, αναφανδόν κατά και τώρα καταπολεμάτε την τρομοκρατία καταπολεμώντας τις μονοπρόσωπες επιχειρήσεις. Δεν ξέρω, ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει κάποια ενδιαφέρουσα απάντηση σε αυτή τη συζήτηση. στις ε, συζητήσεις μας για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στην Ευρώπη ε, και οι φίλοι μας από την αριστερά ε, αυτή τη στιγμή, ενώ αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, δημιουργούν νέα εμπόδια για επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν προκύπτει και μια ευκαιρία που θα μπορούσε να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους, να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ε, ακούμε ένα ε, απόλυτο όχι από την αριστερά. Η δουλειά μας είναι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Αυτές οι μονοπρόσωπες εταιρείες θα υπόκεινται στους ίδιους ελέγχους ακριβώς ε, στους οποίους υπόκεινται και οι υπόλοιπε και από τις αρχές και από την εισαγγελία και από την εφορία. Επομένως ποιος είναι ο κίνδυνος ε, για αυτές τις επιχειρήσεις για την αγορά γιατί πραγματικά εγώ δεν μπορώ να βρω καμία αιτιολογία για τις ανησυχίες σας. Οποιαδήποτε ε, αιτιολογία. Ιδίω ε, το γεγονός ότι ξαφνικά οι απαταιώνες θα βρούνε παραθυράκια για να μπορέσουν να διεξάγουν τις παράνομες δραστηριότητές τους. Τα επίπεδα ελέγχου θα είναι ακριβώς τα ίδια. Αν θέλει κάποιος να ζει ως εγκληματίας, ο οποίος ε, αγνοεί τα διαθέσιμα εργαλεία, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι εγκληματίας και με οποιαδήποτε άλλη μορφή επιχείρησης. Και στην αρχή τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα γιατί δεν μας αφήσατε καμία ευκαιρία να το συζητήσουμε. Την απολαμβάνω βέβαια τη συζήτηση τώρα γιατί καταφέρνουμε και μιλάμε. Θα μπορούσα ίσως να ακούσω και για ποιο λόγο προέκυψε αυτή η ιδέα. Δεν νομίζω ότι ήρθε έτσι καθόντουσαν μια μέρα και δεν είχαν τι να κάνουν. Ε, ε, ε, Υπάρχουν κάποια σημεία που χρειάζονται λίγο βελτίωση και εξορθολογισμό, αλλά δεν μπορεί να λέμε ότι είναι μια περιττή ιδέα που μόνο κακό θα κάνει. Έχω και εγώ συναντηθεί με εκπροσώπους των συνδικάτων και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αυτή η σύσταση μιας μονοπρόσωπης επιχείρησης είναι κάτι το οποίο ε, είναι πολύ γνωστό και δεν δημιουργεί ε, απαραίτητα ε, παράνομες δραστηριότητες και συμπεριφορές. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να αναπτύξουμε το μέσο αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Αν αποτύχουμε, αποτύχαμε, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε μια προσπάθεια. Μπορεί να βοηθήσει πολλούς νέους ανθρώπους να ε, βρουν μια διέξοδο στην αγορά εργασίας. Η κυρία Κομοντίνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το εισηγητή για το έργο του, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση αυτή. Αν θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεωρείται ως ένα κοινοβούλιο που γνωρίζει και κατανοεί τις ευκαιρίες που χρειάζονται οι νέοι επιχειρηματίες, οι ερευνητές και οι καινοτόμοι άνθρωποι. Επίσης, ένα κοινοβούλιο που θα μπορεί να εφαρμόζει τις καινοτόμες ιδέες και να τις μετουσιώνει σε νομοθεσία. Νομίζω ότι η κατάχρηση θα υπάρχει πάντοτε, αλλά κατάχρηση δεν προκύπτει από την νομική ε, έννοια του αν θα μπορέσουμε να δώσουμε περιορισμένη ευθύνη σε μονοπρόσωπη επιχείρηση, αλλά εξαρτάται από τις ε, διαδικασίες διασφάλισης που θα εφαρμόσουμε. Άκουσα τις ανησυχίες με προσοχή. Κάποιες σχετίζονταν με την φοροαποφυγή, με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κτλ. Αλλά μήπως θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε αυτά τα ζητήματα να τα χειριζόμαστε και να τα ρυθμίζουμε μέσω άλλων νομοθετημάτων. Μη, αν είμαστε ε, ε, δυσαρεστημένοι από την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Η λύση δεν είναι να δημιουργήσουμε επιπλέον εμπόδια σε νέους επιχειρηματίες. Επίσης, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν ήδη κάνει το συγκεκριμένο βήμα. Κάποια κράτη-μέλη έχουν ήδη προχωρήσει στο να δώσουν την ε, δυνατότητα σε μεμονωμένα άτομα να μπορούν να συστήσουν ε, μονοπρόσωπες επιχειρήσεις ε, περιορισμένης ευθύνης προκειμένου να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν στην ε, ευρωπαϊκή αγορά. Από αυτή την άποψη η μορφή αυτή της, της, αυτή της επιχείρησης αποτελεί απλώς ένα όχημα και το ερώτημα είναι θέλουμε να δώσουμε περιορισμένη ευθύνη σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Αν η, απο, η απάντηση είναι ναι τότε δεν προκύπτει ότι του δίνουμε αυτομάτως την άδεια να καταφεύγει σε φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία ή να ε, μεταχειρίζεται άσχημα τους υπαλλήλους του. Πρέπει να ε, αντιθέτως ε, φωτίσουμε τις πλευρές που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμογή μιας τέτοιας νομικρής ε, πράξεις. Και νομίζω ότι σε αυτό το δεύτερο έγγραφο που έχει υποβάλει ο εισηγητής υπάρχουν στοιχεία για το πώς θα μπορούσε το συγκεκριμένο εμπορικό όχημα να τύχει της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης. Ο κύριος Ράνιεφ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για τις ε, προσπάθειες που έχει καταβάλει γιατί πρόκειται πραγματικά για μια πολύ δύσκολη έκθεση. Το έγγραφο εργασίας που μας παρουσίασε περιέχει περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδε που απαντούν και στι ανησυχίε που εκφράστηκαν. Θεωρώ ότι η σύνδεση είναι ε, ορθή. Όταν κανείς συνδέει την επιχειρηματική δραστηριότητα με την έδρα, τότε καλύπτει κατά 90% της ισχύουσας νομοθεσίας στο κράτος μέλος. Αυτό που θα ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αν ε, επιτρέπαμε εμπορικούς αντιπροσώπους να έχουν εμπορικές δραστηριότητες σε άλλες χώρες. Οι ανησυχίες ότι η καταχώρηση μέσω ίντερνετ θα μπορούσε να προκαλέσει κατάχρηση, θα σας πω ότι σε 13 ε, κράτη-μέλη υπάρχει αυτή η διαδικτυακή καταχώρηση ε, εδώ και πολλά χρόνια. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα από τη χώρα μου. Πριν από 10 χρόνια είχαμε αυτή τη συζήτηση στη χώρα μου ε, και με τις ίδιες ανησυχίες να εκφράζονται ότι ενδεχομένως να δημιουργηθούν προβλήματα, απάτη, φοροδιαφυγή κτλ. Όμως κάτι τέτοιο ε, δεν επιβεβαιώθηκε στην πραγματικότητα. Αντιθέτως στην χώρα μου ο μόνος τρόπος για να ε, ξεκινήσει κανείς την επαγγελματική του δραστηριότητα είναι μέσω ε, ίντερνετ. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Ας δώσουμε επιτέλους τη δυνατότητα στις μικρές επιχειρήσεις να εργαστούν, να δραστηριοποιηθούν και να μην χρειάζεται να το κάνουν αυτό μέσω εμπορικών αντιπροσωπιών που δεν χαρακτηρίζονται από σταθερότητα, αλλά μέσω εταιριών αυτής της μορφής, εκείνης της μορφής, που θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την μακροχρόνια δραστηριότητά τους και ε, ακολούθως βεβαίως και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Κύριος Κέσνερ, συμφωνώ με πολλούς από όσους έχουν ήδη λάβει το λόγο. Έχω την εντύπωση, εν μέρη τουλάχιστον, ότι προσπαθούν κάποιες πλευρές να μας πείσουν ότι η ίδρυση τέτοιων μονοπρόσωπων εταιρεών είναι πανάκια για να ε, αντιμετωπιστεί η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ αντιθέτως θα έλεγα ωστόσο ότι η ίδρυση μιας τέτοιας μονοπρόσωπης εταιρείας ενδεχομένως να ενέχει και κινδύνους για έναν ε, άνεργο. Το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι όχι η έλλειψη νομοθετημάτων, αλλά η χαμηλή ζήτηση. Αν μάλιστα τώρα στην ανεργία ενός ανθρώπου προσθεθεί και ο κίνδυνος της υπερχρέωσης, τότε έχουμε πρόβλημα. Εμείς θέλουμε βεβαίως να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση, αλλά ε, δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε σε εσφαλμένες υποθέσεις ότι αυτό θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη. Και γι' αυτό το λόγο θα έλεγα ότι ε, οι ισχύουσες διαδικασίες που προβλέπονται για την ίδρυση εταιρείας, εταιρείας είναι χρήσιμες Ακριβώς διότι συνιστούν ένα εμπόδιο το οποίο θα πρέπει να ξεπεράσει κανείς προκειμένου να μπορεί και να διαπιστώσει αν όντω τον συμφέρει ή έχει τη δυνατότητα να ε, γίνει αυτοαπασχολούμενος. Επίσης υπάρχουν και κάποιες ασάφειες στο έγγραφο εργασίας με τις οποίες εμείς ως σοσιαλιστές ε, διαφωνούμε. Εμείς υποστηρίζουμε βεβαίως την ε, αυτοπρόσωπη παρουσία όταν ιδρύεται μια εταιρεία και το ίδιο ισχύει και για το κεφάλαιο ε, που σχετίζεται με τη δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης ε, επιχείρησης με αρχικό κεφάλαιο του 1 ευρώ. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ενέχει πολλούς κινδύνους και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ε, δεν θα πρέπει να υποστηρίξουμε το συγκεκριμένη, τη συγκεκριμένη πρόταση ακριβώς γιατί οι SUP ε, παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον δυναμικό και δεν θα πρέπει να το καταστρέψουμε. Ο Πρόεδρος. Έχει ζητήσει το λόγο η Κομισιόν. Κύριε Χόγκερ, πολύ σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λεγκράντε για τον εισηγητή, για το επίμονο έργο του και για τη διάθεσή του να ε, εξευρεθεί συμβιβαστική λύση και να ληφθούν υπόψη και οι απόψεις των ε, ε, πλέον επιφυλακτικών ευρωβουλευτών. Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο για την διευκόλυνση των μικρομεσών επιχειρήσεων. Ξέρουμε ότι οι συζητήσεις στο Κοινοβούλιο ήταν δύσκολες και εμείς εξακολουθούμε να αξιολογούμε το συγκεκριμένο κείμενο, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Ε, βλέπουμε ότι ο εισηγητής έχει κάνει κάποιες προτάσεις για να διασκεδαστούν οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί. Ε, και αυτές επικεντρώνονται γύρω από το ζήτημα του κινδύνου της κατάχρησης του νομοθετήματος. Και ποιος δεν θα ήθελε άλλωστε. Ε, ένας από τους τρόπους βεβαίως είναι ο περιορισμός του πεδίου ισχύου, του πεδίου για τις μικρές ή πολύ μικρές εταιρείες. Αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες καινοτόμες ιδέες όπως το κριτήριο της οικονομικής δραστηριότητας που εισάγεται στο κείμενο του συγητή. Υπάρχει η απέτηση ε, ότι κάθε εταιρεία που θέλει να υπαχθεί σε αυτό το καθεστώ θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι έχει ένα χρόνο ε, ε, εμπορική οικονομική δραστηριότητα στον συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, αν δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, υπάρχει πρόβληση για το πώς μπορεί να διαλυθεί μια τέτοια εταιρεία. Επίσης, πιστεύουμε ότι η συγκητής έχει ε, καταδείξει ε, πιθανές λύσεις που θα μπορούσαν να επιλεγούν και ελπίζουμε ε, ότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους ευρωβουλευτές να συζητήσουν πιο ενεργά, ε, να συμμετάσχουν πιο ενεργά σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι επικεντρωνόμαστε ίσως λίγο υπερβολικά πολύ στο 0, κάτι της της απάτης και ξεχνούμε μάλλον το 99,9% ε, των ε, υγιών εταιριών που δεν καταφεύγουν σε απάτες. Και όπως υπόθηκα, υπόθηκε και ε, από άλλους, το εργαλείο αυτό, ο μηχανισμός αυτός έχει ζητηθεί από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. Εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας για να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα και για να διασκεδάσουμε και τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί στη διάρκεια της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντεγκράντες, πολύ σύντομα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ την Κομισιόν για τις αξιολογήσεις της. Γνωρίζαμε ήδη ότι ε, το να είναι η νέα έδρα και παρά το γεγονός ότι ε, υπήρχε δυσκολία στη μετάφραση, μεταφράστηκε πάρα πολύ σωστά. Δεν υπάρχει ε, καμία αμφιβολία για μένα ότι η διοικητική έδρα είναι η ίδια. Επιπλέον, εγώ ε, παραδέχομαι ότι ίσως είναι μια υπερβολή της οδηγίας, αλλά δεν έχουμε χρόνο, αλλά αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από νομική σκοπιάς. Έπρεπε να γίνει κανονισμός ή οδηγία. Γιατί έκανε οδηγία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ο κανονισμός απέτυχε ε, και επομένως χρειαζόταν μια ευρύτερη πρόταση. Η οδηγία περιλαμβάνει μεγαλύτερη ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν με ευελιξία αφενός να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν όπως νομίζω ότι άλλωστε ότι φαίνεται σαφέστατα στο έγγραφο εργασίας ε, που σας παρουσίασα, αλλά ταυτόχρονα διαπίστωσα ότι αυτό ε, δημιουργεί αμφιβολίες όχι στον κανονισμό, ναι στην οδηγία και ναι στην ευελιξία, αλλά αμφιβολίες για το κατά πόσον αυτό μπορεί να δημιουργήσει σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Ε, σίγουρα δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση αυτή είναι σαφέστατα ιδεολογικού χαρακτήρα και προκύπτει ως συνέπεια μιας νέας κατάστασης στην Ευρώπη και στον κόσμο. Υπάρχουν κάποια προβλήματα ε, διαρθρωτικής ανεργίας, ε, έρχονται τα ρομπότ και αφαιρούν τις θέσεις εργασίας από τους ε, ανθρώπους και υπάρχουν κάποιες παραδόσεις σε κάποιες χώρες, αυτό το, το παραδέχομαι, αλλά αυτό είναι ε, απαρχαιωμένες αντιλήψεις. Και πιστεύω ότι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας δεν γίνεται να δημιουργηθεί από την ακαμψία των παλιών εργασιακών μοντέλων, θα γίνει στον νέο ψηφιακό κόσμο και οι νέοι μας ζητούν να περάσουν από την επελπισία και την ανεργία στην αυτοαποσχόληση και το προσπαθεί όλος ο κόσμος και χρειάζονται ένα εργαλείο. Μπορεί ίσως να μην είναι επαρκώς ευφυές ή επαρκές ή να περιλαμβάνει κινδύνους, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι ε, ε, εξαφανίστηκαν κάποιες μορφές απασχόλησης ε, και υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ήταν απόλυτα προετοιμασμένοι για να ακολουθήσουν νέες ε, μορφές εργασίας. Και επομένως ε, ε, οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να εργαστούν και λένε ναι. Αλλά βλέπω ότι από πολιτική σκοπιά η πρόταση αυτή, πέραν της προσπάθειας που έκανα να αποδεχτώ όλες τις ανησυχίες από όλες τις πλευρές, γιατί θεωρώ ότι λογικά υπάρχουν ανησυχίες, φαίνεται ότι τη βλέπουν όλοι αρνητικά γιατί δεν θέλουν να προχωρήσει η πρόταση. Θα είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να επιβιώσει αυτή η πρόταση. Αλλά σήμερα πρέπει να σας πω ότι εδώ δεν άκουσα κάποιες νέες θέσεις ή κάποια επιχειρήματα σε σχέση με τα προηγούμενα που ακούσαμε την πρώτη φορά, όταν όντως ε, το προηγούμενο έγγραφο εργασίας περιλαμβάνει πάρα πολλές ε, ρήτρες ασφαλείας για να μπορέσει να διαφυλάξει κάποια πράγματα και ε, να μην υπήρχαν και στο προηγούμενο που δεν υπήρχαν. Τώρα, θέλετε ή δεν θέλετε. Εγώ δεν ξέρω αν η συζήτηση αυτή είναι προοδευτική. Σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες. Ε, μήπως αυτό σημαίνει απλώς και ε, απομόνωση και ακαμψία και ε, φόβο απέναντι στα νέα μοντέλα το είπα και στην αρχή, ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι ίσως πιο φιλόδοξη και να κάνει ένα, μοντέλο, ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικής ε, ε, νομοθεσίας. Ε, αυτά μπορούν να τα διορθώσουμε μέσω ευελιξίας, αλλά να πάμε παραπέρα δεν γίνεται. κύριε Πρόεδρε, εγώ προσπάθησα να κάνω μία τελευταία προσπάθεια θα μιλήσουμε σοβαρά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα καταλήξουμε και σε κάποια απόφαση, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αναγνωρίζετε την προσπάθειά μου και σας διαβεβαιώ ότι πραγματικά προσπάθησα και το ξέρετε ότι προσπάθησα. Και όχι επειδή είναι ε, παιδί μου αυτή η έκθεση, γιατί δεν είναι, Τη Κομισιόν είναι το τέκνο. Επομένως, εμείς θέλαμε απλώς να το συνοδεύσουμε και μέσω της κατάλληλης διαδικασίας να γίνει ίσως ε, ε, αποδεκτό για, με έναν ελάχιστο παρονομαστή. Μετά από αυτά που άκουσα βέβαια έχω πραγματικά αμφιβολίες και βλέπω ότι υπάρχουν πολλές άκαμπτες θέσεις. Και αυτά είναι τα πράγματα, έτσι έχουν τα πράγματα κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ε, εκτιμώ τα όσα άκουσα, δεν άκουσα κάτι καινούριο στις ενστάσεις σας. Ε, η ε, συνάδελφος Ευρωβουλευτής από τη Σουηδία αναφέρθηκε σε κάποιες εκθέσεις για τους κινδύνους και αναφέρθηκε στην τρομοκρατία. Πραγματικά νομίζω ότι υπερβάλλουμε εδώ ε, και δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες εξέδωσαν ένα τέτοιο έγγραφο. μου φαίνεται υπερβολή χωρίς καμία αμφιβολία γιατί δεν ισχύει και πραγματικά δεν είναι αλήθεια ότι αυτό προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για απάτη, για έλλειψη εγγύησεων εάν χρησιμοποιηθεί. Πρόκειται για ένα κίνδυνο τον οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε πολλές περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από αυτά που άκουσα σήμερα και από τις ερωτήσεις που έχουν διατυπώσει και κάποιοι που είναι απόντες, ε, ε, ε, διότι δεν είναι όλοι εδώ, είναι, είναι πέμπτη απόγευμα που όλοι φεύγουν και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε μια έκθεση για να ακολουθήσουμε τη συνήθιση διαδικασία ή να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να λάβει μια απόφαση προς την αντίθετη κατεύθυνση και να μπορέσει ίσως να αλλάξει και στάση για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you Και εμείς σας ευχαριστούμε. Μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο της σημερινής διάταξης. Είχαμε συμφωνήσει ότι θα συζητήσουμε τα σημεία 16 και 17 της της διάταξης. Και μετά σας προτείνω να αναβάλουμε τη συζήτηση για το 14 και το 15, γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε με την συνεδρία κυκλισμένων των θυρών. ότι υπάρχει μια υπόθεση άρσης ασυλίας που πρέπει να συζητηθεί σήμερα, γιατί αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει γέρος. Ε, επίσης ζητώ ησυχία στην αίθουσα. Uh, thank you. Uh, Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, το σημείο 16 και το 17 Φορούν στην υπογραφή και επικύρωση εκ μέρου των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you very much for silence. Σας ευχαριστώ που κάνετε ησυχία. Θέλω να ξεχωρίσουμε ε, ακριβώς ε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του 16 και του 17. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για τη δικαστική συνεργασία σε αστικέ υποθέσεις, στο πρώτο σημείο, ενώ στο δεύτερο είναι το πρωτόκολλο ως προ τα υπόλοιπα στοιχεία με την εξαίρεση των πτυχών δικαστική συνεργασίας σε αστικέ υποθέσεις. Είναι λοιπόν το, η Διεθνής Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη και την Αποζημίωση σε συνδυασμό με την μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών στην θάλασσα, διαθαλάσσης. Είναι μια σύμβαση η οποία πρέπει να επικυρωθεί ακόμα και από άλλα κράτη πριν να τεθεί σε ισχύ μια και στο κείμενο του ούτε τη σύμβαση ούτε του πρωτοκόλου δεν υπάρχει κάποια ρήτρα για την σύναψη για τη δυνατότητα μάλλον να είναι συμβαλόμενο μέρος κάποιο περιφερειακό οικονομικός, ε, οργαν, κάποιος οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν την επικύρωση. Αυτό γίνεται μετά από ε, πρόταση της Επιτροπής ε, θετική γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απόφαση του Συμβουλίου με βάση το άρθρο 218 παράγραφος 6 σημείο α της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, στις 10 Δεκεμβρίου 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έδωσε τη συγκατάθεσή του στο προσχέδιο της ε, απόφασης του Συμβουλίου. Ωστόσο, οι αποφάσεις τις οποίες ενέκρινε το Συμβούλιο ε, αποκλίνουν σε σημαντικό βαθμό ε, από την πρόταση της Επιτροπής ως προς τα εξής. Πρώτα απ' όλα, με βάση όσον αφορά μάλλον το πεδίο όπου αναγνωρίζεται αποκλειστική αρμοδιότητα με βάση το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γεγονό ότι εδώ υπάρχει μια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ του πεδίου εφαρμογή τη σύμβαση αυτή και τη οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη. Δεύτερον, χρειάζεται ένα ε, να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την επικύρωση από το, του πρωτοκόλλου αυτού έτσι ώστε να μην υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού και ιδιαίτερα ε, πλέον εκτίματα που θα μπορούσαν κάποιοι οικονομικοί παράγοντες, και ε, κάποιες επιχειρήσεις να έχουν. Τρίτον, ποια είναι η κατάλληλη νομική βάση της ε, απόφασης του Συμβουλίου. Το άρθρο 192 της Συνθήκης για τη Λειτουργία που αναφέρεται στην αστική ευθύνη σε περίπτωση ε, περιβαλλοντικών καταστροφών ή το άρθρο 100 ε, παράγραφος 2 που σε συνδυασμό με το 218 παράγραφος 6 για τις μεταφορές. Και στις δύο περιπτώσεις δηλαδή 100 παράγραφος 2 και 192 του ε, ε, ε Σύμβαση για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις δύο λοιπόν αυτές περιπτώσεις περιπτώσει εφαρμόζεται η συνήθι ε, νομοθετική διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και ο διαρκής εισηγητής για θέματα νομικής βάσης ο κ. Άξελ Βος θα μπορούσε με δικιά της πρωτοβουλία να εφαρμόσει τον κανόνα 39 του κανονισμού και να εξετάσει κατά πόσο αυτή η αλλαγή στη νομική βάση που έγινε δικαιολογείται. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στην Επιτροπή και μετά στο Συμβούλιο για να μας εκφράσουν τις θέσεις τους για τα θέματα αυτά. Η Επιτροπή πρώτη. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη γιατί αναφερθήκατε ήδη περιληπτικά στα τρία ε, σημεία στα οποία η Επιτροπή και το Συμβούλιο διαφωνούν. Ένα από αυτά αναφέρεται μόνο στο πρωτόκολλο που ε, σχετίζεται με την καθιστική συνεργασία και ξεκινώ λοιπόν με την αλλαγή της νομικής βάσης. Ε, η αλλαγή που έγινε από το 192 και το 100 παράγραφος 2. Αυτό ε, παραγνωρίζει μια πολύ βασική πρόνοια του ε, συμφώνου του 2016 ε, για τη μεταφορά αυτών των βλαπτικών ουσιών που είναι η αρχή ότι ο, ο ρηπαίνων πληρώνει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι είναι, εφαρμόζεται και σχετίζεται αυτό το πρωτόκολλο με την οδηγία για τις, την περιβαλλοντική αστική ευθύνη. Εάν δεν βασιστούμε στη νομική βάση που συμπεριλαμβάνει και αυτά, ε, στην πραγματικότητα υπονομεύουμε ένας από τους βασικούς στόχους ύπαρξης αυτούς της ε, σύμβασης του 2010, δηλαδή να πάψει να υπάρξει, ε, υπάρχουν περιστατικά σοβαρή ρήπανση στη θάλασσα. Γνωρίζετε ότι όταν επικαιρώνεται μια διεθνή συνθήκη εξετάζεται ποια είναι η βασική στόχευση αυτή τη διεθνού συνθήκη για να αποφασιστεί και ποια είναι η κατάλληλη νομική βάση η Επιτροπή διαφωνεί με την αξιολόγηση που κάνει το Συμβούλιο ως το ποια είναι η κατάλληλη νομική βάση εδώ. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της αποκλειστικής αρμοδιότητας, η θέση της Επιτροπής είναι η εξής. Η εφαρμογή του Συμφώνου του 2010 είναι ε, πλήρης, εφαρμόζεται σε μια σειρά κανόνων και δεν μπορεί να, ε, να περιοριστεί σε ένα μέρος των ε, προνοιών του συμφώνου. Για αυτόν τον λόγο θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ευρεία ερμηνεία. Επίσης, δεδομένου ότι τα κράτη-μέλη ασκούν τη δικιά τους αρμοδιότητα είτε όταν δεν ασκεί αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιλέξει έχει αποφασίσει να μην ασκήσει αρμοδιότητες που τις αποδίδονται από τη συνθήκη ε, και δεδομένων των προβλέψεων της οδηγίας για το περιβάλλον θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτή η αποκλειστική αρμοδιότητα στην εφαρμογή του Συμφώνου του 2010. Επίσης, διαφωνούμε με την αλλαγή που έγινε σε σχέση με το άρθρο 100 παράγραφος 2, γιατί εδώ πλέον Δεν ζητείται από τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν το σύμφωνο ε, έχοντας την υποχρέωση αποτελέσματος να, να, το πράξουν, αλλά μόνο να ε, το επιδιώξουν. Ε, επί τη βάση της ε, ορθής συνεργασίας προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν οποιοδήποτε μέτρο, είτε γενικό είτε ειδικό, για την ε, εφαρμογή των προβλέψεων της συνθήκης ή του παράγωγου δικαίου. Επίσης, για πρακτικούς λόγους θέλω να επισημάνω κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι προκειμένου, ε, εάν μάλλον το σύμφωνο επικυρωθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ομοιόμορφα και από όλου, αυτό διασφαλίζει την ισότητα και τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού, κάτι που είναι και στόχο του, του Συμφώνου και του Πρωτοκόλλου του 2010. Εάν πάμε σε μια κατάσταση όπου κάποια κρατημέλη θα έχουν επικυρώσει το σύμφωνο του 2010, ενώ άλλα θα ε, ακολουθούν τις πρόνοιες της ε... ε... οδηγίας της περιβαλλοντικής της Ένωσης, αυτό σημαίνει ότι ε, θα μπορεί ε, ο πλειοκτήτης να επιλέξει την πιο ευνοϊκή για αυτόν νομοθεσία κάτι το οποίο θα μπορούσε επίσης να πλήξει δυσμενώς και τα θύματα σε περίπτωση περιβαλλοντικής καταστροφής στη θάλασσα. Η Επιτροπή διαφωνεί λοιπόν με αυτήν την πολιτική, με αυτήν την, ε, την α, πιθανότητα. Σας ευχαριστώ. Το Συμβούλιο, παρακαλώ, έχει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Το πρωτόκολλο HNS είναι σημαντικό για να ολοκληρωθεί το διεθνές νομικό πλαίσιο για την αστική ευθύνη και την αποζημίωση που σε περίπτωση πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπους και στο περιβάλλον. Πολλά κράτη-μέλη είναι έτοιμα να κυρώσουν την ε, συγκεκριμένη σύμβαση και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε μια εξοδότηση ταχεία για να προχωρήσουν σε αυτήν την ενέργεια. Για την νομική βάση, το Συμβούλιο ε, προτείνει την αλλαγή της νομικής βάσης από περιβάλλον σε μεταφορές, διότι δεν αφορά το ζήτημα μόνο το περιβάλλον, αλλά αφορά και εκρήξεις ή ε, φθορές σε περιουσιακά στοιχεία ή ε, θανάτους ανθρώπων που σχετίζονται και με τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με την ε, οδηγία ε, τη σχετική του ε, Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στόχος είναι να υπάρχει προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών επικίνδυνων ουσιών. Ωστόσο αυτό δεν αφορά τους τραυματισμούς ή την φθορά περιουσίας. Ε, το ζήτημα αυτής της οδηγίας και του πρωτοκόλλου HNS καλύπτονται σε ένα βαθμό αλλά δεν ταυτίζονται. Γι' αυτό το λόγο το Συμβούλιο ζητά να διατηρήσει την αρμοδιότητα όσον αφορά το πρωτόκολλο στο βαθμό που δεν αφορά κοινούς κανόνες. Όσον αφορά την δικαστική συνεργασία, το Συμβούλιο θεωρεί ότι τα άρθρα 37, 41 και 43 του κεφαλαίου 1 του πρωτοκόλου HNS δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι παραπομπές σε αυτά τα άρθρα που ε, είναι μόνο βοηθητικά προς τις ε, κύριες διατάξεις θα πρέπει να διαγραφούν από την πρόταση της Κομισιόν. Και όσον αφορά την κύρωση, το Σύμβουλο το Συμβούλιο δεν μπορεί να δεχτεί ε, υποχρέωση κύρωσης εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει ε, προταθεί από την Κομισιόν. Χρειαζόμαστε ευελιξία προκειμένου να μπορέσουν τα κράτη-μέλη που θέλουν να κυρώσουν το πρωτόκολλο να το κάνουν όσο το δυνατόν συντομότερο χωρίς να ε, καθυστερούνται από άλλα κράτη-μέλη που χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Ωστόσο υπάρχει ευρεία ε, συνένεση στο Συμβούλιο ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστεί δυνατή η κύρωση του πρωτοκόλλου το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, δεν βλέπω κάποιος άλλος να ζητά το λόγο. Με την άδειά σας λοιπόν θα ήθελα ε, τον ε, μόνιμο εισηγητή μας για την νομική βάση, τον κύριο Άξελ να μας δώσει να μας παρουσιάσει την άποψή του και θα προχωρήσουμε αργότερα στην συζήτηση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση. Επίσης, με την άδειά σας θα αναβάλουμε τη συζήτηση των σημείων 14 και 15 και θα προχωρήσουμε στην συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών. Επομένως, θα ήθελα να ζητήσω ε, να εγκαταλείψουν την αίθουσα όσοι δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί